Καλησπέρα σας κυρίες, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας εύχομαι ένα θερμό καλωσόρισμα στη σημερινή συνεδρίαση. Έχουμε πολλά σημεία στην ημερήσια διάταξη και ελπίζω όλοι να λάβετε γνώση ότι θα συζητήσουμε κάπως αργότερα την έκθεση Στρέλα αλλά θα αρχίσουμε με ένα ενημερωτικό σημείωμα τις χθεσινές αποφάσεις της συνεδρίασης των συντονιστών. Αποφασίσαμε να καταρτήσουμε τρεις εκθέσεις πρωτοβουλίας. Η πρώτη αφορά το μέλλον των κοινοφελών υπηρεσιών, των υπηρεσιών ε, γενικού ενδιαφέροντος. Θα την αναλάβουν οι φιλελεύθεροι. Η δεύτερη έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας αφορά τις δημογραφικές προκλήσεις και την ε, αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Θα τη συντάξει το ΕΛΚ. Και η τρίτη έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας που λέγεται, φέρει τον τίτλο «Ανάπτυξη του δυναμικού απασχόλησης σε μια νέα αηφόρο οικονομία» Ε, δόθηκε στους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Οι συντονιστές έλαβαν απόφαση και για την ακρόαση με τίτλο «Προς μία νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων». Αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε έξι εμπειρογνώμονες στη δημόσια αυτή ακρόαση. Θα σας διαβάσω τα ονόματά τους κυρία, η κυρία Νταρμόλιν, κυρία Βάλμπη, κυρία Βασιλιάδου, κυρία Σονέτο, η κυρία Φελίπε, και θα προσκαλέσουμε και έναν εμπειρογνώμονα από τη Βουλγαρία, αλλά περιμένουμε ε, τους φιλελεύθερους να μας κοινοποιήσουν το όνομά του ή της. Θα προβλέψουμε και δύο αναπληρωτές αν κάποιος ε, από τους εμπειρογνωμονές μας ε, δεν καταφέρει να παραστεί στη δημόσια ακρόαση. Και αποφασίσαμε και ποια θα είναι τα μέλη του, τα μέλη του πάνελ αυτής της ακρόασης. Ο εισηγητής και ο σκιώδης εισηγητής αρμόδιοι για τα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τη Διεθνή ημέρα της γυναίκας, που θα εορταστεί με εκδηλώσεις 16 Μαρτίου αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με τις ε, Επιτροπές Ανάπτυξης ε, την Νομική Επιτροπή, θα προσκαλέσουμε τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κάποιον από το UNIFAM και εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας. Επίσης θα προσκαλέσουμε και διάφορες οργανώσεις που έχουν εκπονήσει ενδιαφέρουσες μελέτες. Για παράδειγμα το Ίδρυμα του Δουβλίνου που έχει καταρτήσει μελέτες για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των βιωτικών συνθήκων. Επίσης θα προσκαλέσουμε εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών, την κυρία Εύα Ένσλερ, συγγραφέα μεταξύ άλλων και τον μονολόγο του Εδίου. Επίσης ε, θα μιλήσουμε και για τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως το διαδικτύο, το facebook και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο. Αυτή είναι η βασική διάρθρωση της ε, εκδήλωση που θα γίνει στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και θα ενημερωθείτε για την πορεία των προετοιμασιών. Επόμενο σημείο, το πρόγραμμα εργασιών για το 2010. Οι συντονιστές αποφάσισαν να αναθέσουν ε, τη σύνταξη δύο μελετών ε, σε επιρρογραμμόνες, για παράδειγμα τη χρηματοπιστωτική κρίση και τις συνέπειές της ε, στις θέσεις εργασίας των γυναικών, καθώς και το σχετισμό με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια του για να προωθήσουν ε, θέσεις εργασίας για τις γυναίκες. Επίσης, ε, θα ζητήσουμε την εκπόνηση μελέτης για το κοινωνικό δίκτυο ασφάλειας για τις εγγύους και αυτές ήταν ολίγης οι αποφάσεις που έλαβαν χθες οι συντονιστές. Συζητήσαμε και λάβαμε απόφαση για το πώς ε, θα διαχειριστούμε τα νέα θέματα της διαδικασίας συναπόφασης. Ιδιαίτερα όταν ε, θα τροποποιηθούν και θα ενισχυθούν και οι εξουσίες των Εθνικών Κοινοβουλίων στα πλαίσια της διαδικασίας της επικουρικότητας. Τα πρακτικά φυσικά θα μοιράσουμε από τη χθεσινή μας συνεδρίαση σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Και ερχόμαστε στο σημείο 10. που θα μετατοπιστεί προς το τέλος της σημερινής ε, ημερήσιας διάταξης ε, το θέμα της αποστολής μας στη Μαδρίτη θα το αφήσουμε τελευταίο και θα περάσουμε στο 11 προς το παρόν τις πτυχές που αφορούν το φύλλο σε εκθέσεις προόδου 2009 για την Κροατία, την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Τουρκία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εμείς θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του ψηφίσματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τη διεύρυνση, στην έκθεση πρόοδου δηλαδή. Και γι' αυτό, για να κάνουμε πιο αισθητή την συνεισφορά μας, αποφασίσαμε να καταθέσουμε τροπολογίες που θα συμπεριληφθούν στο ψήφισμά μας που θα υποβάλουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών. Αν εγκρίνουμε αυτό το ψήφισμα σήμερα, θα το υποβάλουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών. Θα το υποβάλει ο Πρόεδρος εκ μέρους της Επιτροπής και θα το υποβάλουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών από κοινού. Εγώ με τα μέλη της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων της Γυναίκας που είναι μέλη και της Επιτροπής Εξωτερικών. Το ψήφισμά μας απαρτίζεται από πολλές παραγράφους Δύο αναφέρονται στην Κροατία. Εκεί τονίζουμε τη σημασία που έχει η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και η ανάγκη πάταξης των διακρίσεων κατά των γυναικών σε ό,τι αφορά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Επικροτούμε το γεγονός ότι υπάρχει ε, μια γενική ευαισθητοποίηση για το θέμα της κακοποίησης των γυναικών, της βίας κατά των γυναικών. Και τονίζουμε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ε, κυρίως ε, για παροχή συνδρομής προς τα θύματα αυτής της βίας. Για την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, χαιρετίζουμε τη νέα νομοθεσία που κατοχυρώνει ισότητα ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων και σημειώνουμε ότι παρόλο που υπάρχει ακόμη μίζον πρόβλημα με τη βία κατά των γυναικών η νομοθεσία τουλάχιστον κατοχυρώνει με προστασία των γυναικών, αλλά φυσικά δεν χρειάζεται μόνο νομοθεσία στα χαρτιά, χρειάζεται και έμπρακτη εφαρμογή της. Για την Τουρκία αναγνωρίζουμε ε, την ύπαρξη νομικού πλαισίου για την απαγόρευση της βίας κατά των γυναικών και των καταναγκαστικών γάμων, αλλά εντοπίζουμε κάποιες αδυναμίες και κενά στην εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Τέλος, να πιστούμε την προσοχή στο γεγονό ότι το επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας της Τουρκίας είναι από τα χαμηλότερα μεταξύ των χωρών ΟΣΑ. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για να εισέλθουν οι γυναίκες στην αγορά και να εξασφαλίσουν μια οικονομική ανεξαρτησία. Αυτά με λίγα λόγια πραγματεύονται οι τροπολογίες που ψηφίζουμε, που θα εγκρίνουμε, αφού τις συζητήσουμε βέβαια. Η ε, κυρία Κορνέλησε ζήτησε πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής Έχουμε κάποιες ε, τροπολογίες που θα καταθέσουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για αυτά τα θέματα. Και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία τα εξετάζουν και διαφορετικές επιτροπές σε αυτό το κοινοβούλιο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε επί του επιστήτου, αλλά πρέπει να προβάλλουμε ποια είναι η γενική προσέγγιση και τι είναι σημαντικό όταν καταθέτουμε τροπολογίες. Εμείς ως μέλη της Επιτροπής Γυναικών, προφανώς είμαστε μέλη και σε άλλες επιτροπές και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της διάστασης του φίλου που έχουμε στα χέρια μας. Εμείς οι ίδιες με το να συμμετέχουμε και αλλού αποδεικνύουμε στην πράξη τη διάσταση του φύλου. Το θέμα είναι τι αναφέρεται στις εκθέσεις πρόοδου αυτών των χωρών. Ω συντονίστρια και ω μέλο Επιτροπής Επιτροπή Υποθέσεων, εγώ συνέβαλα στη σύνταξη αυτών των τροπολογιών και ευελπιστώ να τύχουν τις μεγάλες υποστήριξη από την Επιτροπή μας, γιατί αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Ε, ελπίζω όμως ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Και έτσι λοιπόν όπως σας είπα ελπίζω ότι θα συμμετέχουμε έντονα σε πολλές άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζοντας τη διάσταση του φίλου. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κορνέλισεν. Πράγματι, εδώ πρόκειται για μια μέθοδο εργασία που είναι ιδιαίτερα θετική για την Επιτροπή μας, γιατί με τον τρόπο αυτό μας προσφέρονται πολλές ευκαιρίες έτσι ώστε να προβάλλουμε τα δικά μας τα θέματα στις υπόλοιπες επιτροπές. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο, ως εκ τούτου προτείνω να περάσουμε στην ψηφοφορία και προτείνω να ψηφίσουμε και τις επτά τροπολογίες από κοινού στο σύνολό τους. Συμφωνείτε? Ψηφίζουμε λοιπόν. Ε, ποιος είναι παρακαλώ υπέρ, να σηκώσει το χέρι του. Υπέρ του ψηφίσματός μας. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε λοιπόν το ψήφισμά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη πώς μπορούμε ε, να εμποδίσουμε και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την εμπορία ανθρώπων. Πρόκειται εδώ κυρίως για την προστασία των θυμάτων. Το θέμα είναι το εξή. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, που σήμερα θα τεθεί σε ισχύ η εμπορία ανθρώπων πλέον περνάει από τη διαδικασία διαβουλεύσεων στη διαδικασία της ε, συναπόφασης. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο σε αυτά τα θέματα. Η συνθήκη της Λισαβόνας, όταν αυτή θα τεθεί σε ισχύ, αυτό σημαίνει ότι η πρόταση που κατέθεσε η Κομισιόν θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια άλλη πρόταση η αρμόδια κατά κύριο λόγο είναι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και η δική μας Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί με γνωμοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ε, συμφωνήσαμε ε, ο εισηγητής της ΛΥΜΠΕ και η δική μας εισηγήτρια, η κυρία Μπάουα, συμφωνήσαμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή να μην τοποθετηθούμε στην πρόταση που έχει ήδη κατατεθεί γιατί όπως σας είπα θα κατατεθεί νέα πρόταση και θα περιμένουμε μέχρι να έρθει από την Επιτροπή η νέα πρόταση και κατόπιν θα συζητήσουμε το θέμα μέσα στη διαδικασία της συναπόφασης. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, τοποθετηθεί το συντομότερο δυνατόν σε αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα της ε, εμπορίας ανθρώπων, έτσι ώστε οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορούν να συμπεριληφθούν στη νέα πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο εισηγητής ε, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και η δική μας ε, εισηγήτρια για το λόγο αυτό συμφώνησαν να διαμορφώσουν μια προφορική ερώτηση. Κρίναμε ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση εν ώψη της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Εμείς ε, λοιπόν καλούμεθα τώρα να αποφασίσουμε να καταθέσουμε ε, δύο προφορικές ερωτήσεις προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συζητήσαμε λοιπόν για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Είναι πολύ πιθανόν και η Επιτροπή αυτή να ε, διατυπώσει προφορική ερώτηση. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς, πώς εμείς θα διατυπώσουμε τη δική μας. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα συζητήσουμε σήμερα το θέμα αυτό. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπάουα για να μας ε, ενημερώσει που ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτές τις δύο προφορικές ε, ερωτήσεις. Κυρία Μπάουα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που περιγράψατε σωστά την κατάσταση. Το θέμα αυτό καλύπτεται από μια ιδιαίτερη διαδικασία η οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχε και για το λόγο αυτό προκύπτουν αρκετά προβλήματα. Υπάρχουν λοιπόν δύο λύσεις. Η πρόταση κατατέθηκε έγκαιρα στο Κοινοβούλιο για την απόφαση πλαίσιο και εμείς είτε μπορούμε να δεχθούμε τη διαδικασία της συναλλαγής και αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει τις αμέσως επόμενες μέρες να εγκρίνει αυτήν την απόφαση πλαίσιο. Από την άλλη βέβαια είναι σαφές ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ε, θα τεθεί σε ισχύ ως εκ τούτου η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών αλλά και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι πρέπει να προτιμήσουμε τη διαδικασία της συναπόφασης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ενημερώσουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή το ότι είναι σημαντικό για μας και πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτή την απόφαση πλαίσιο. Για το λόγο λοιπόν αυτό επιλέξαμε αυτή τη διαδικασία, αποκοινούμε την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Γνωρίζετε επίσης ότι θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με την ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Η συνεργασία με την κυρία Χέντ ήταν άψογη. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, σε αυτή τη ε, διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα εγκρίνει αυτό το κείμενο. Η διαδικασία είναι, όπως σας είπα και πριν, ασυνήθιστη. Είναι τελείως καινούρια. Και ως εκ τούτου υπάρχουν κάποια προβλήματα στην ε, εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. τα ερωτήματα που έχουν τεθεί έχουν διατυπωθεί πολύ σωστά, αλλά υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, ε, κυρίως ε, εκ μέρους των πρασίνων. <clears throat> Όχι μόνο γιατί η διαδικασία είναι ασυνήθιστη, αλλά και ο τρόπος εργασίας για αυτό το θέμα. Το χρονικό διάστημα ήταν περιορισμένο, γι' αυτό το λόγο συμπεριλάβουμε όλους του ε, σκιώδη και από τις δύο επιτροπές. Ασυνήθιστο και αυτό, αλλά μόνο έτσι ε, μπορέσαμε να επιταχύνουμε λιγάκι τις ε, διαβουλεύσει. Ήθελα επίσης να επισημάνω ότι οι πράσινοι έχουν κάποιες επιφυλάξεις ελπίζω βέβαια οι επιφυλάξεις αυτές να οφείλονται μόνο σε παρεξηγήσεις. υπάρχουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της ζήτησης. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστεί το θέμα της ζήτησης γιατί στην ανάλυση στην οποία έχουμε προβεί διαπιστώνουμε ότι και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και οι εκθέσεις του ε, Διεθνούς ε, Οργανισμού Εργασίας καταλήγουν στο ότι αυτό το φαινόμενο για το οποίο συζητάμε προκύπτει και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζήτηση. Η ζήτηση λοιπόν είναι η κινητήρια δύναμη όλου αυτού. Και γι' αυτό σας εξηγώ ότι συμπεριλάβαμε όλους τους σκιώδης ηγητές, όλοι οι σκιώδης ηγητές συμφώνησαν και θα ήθελα να παρακαλέσω την Κομισιόν να στηρίξει το κείμενό μας Αργότερα θα περάσουμε στο ίδιο το κείμενο της απόφασης που έχει κατατεθεί για να ληφθεί απόφαση. Το κείμενο αυτό είναι μακροσκελές θα έλεγα και έχει και αυτό κάποια προβλήματα. Εγώ θα έλεγα να συμφωνήσουμε στο δικό μας το κείμενο το οποίο κείμενο θα το καταθέσουμε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών και ε, όταν θα το καταθέσουμε θα σας παρακαλέσουμε να το εγκρίνετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφα από τη Γραμματεία, την Κάρολιν, η οποία ε, στάθηκε αρρωγός στην προσπάθειά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Κάρολιν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάουερ. Ήταν ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Έχουμε να κάνουμε με έναν νέο τρόπο εργασίας εδώ, κάπως ιδιαίτερο τρόπο εργασίας και είναι καλό οι σκιώδεις εισηγητές και οι εισηγήτριες εξ αρχής να εμπλέκονται στην προσπάθεια που γίνεται. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Αν όχι μπορούμε νομίζω να κάνουμε δεκτές τις δύο προφορικές ερωτήσεις. Το σημειώνω αυτό και συνεχίζουμε. Προχωράμε. Θα ήθελα να σας προτείνω τώρα να ψηφίσουμε τις δύο προφορικές ερωτήσεις από κοινού. Συμφωνείτε για την κατάθεσή τους, ποιες, ποιες είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εντάξει λοιπόν κλείσαμε και το τυπικό, οι δύο προφορικές ερωτήσεις γίνονται δεκτές και συγχαρητήρια στην κυρία Μπάουα η οποία ολοκλήρωσε σε συνεργασία με την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών την προσπάθεια αυτή. Το επόμενο σημείο στην ημέρηση διάταξη Πρόκειται για το θέμα της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγγύων, λεχόνων κτλ. Να σας θυμίσω εδώ Είχε απορριφθεί στις 9 Μαΐου η έκθεση με την οποία ασχολούμεθα και οι συντονιστές αποφάσισαν να γίνει μια νέα προσπάθεια και έχουμε ορίσει την κυρία Εντίτε Εστρέλα η συγγήτρια. Στις 4 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας κάναμε μια πρώτη συζήτηση με την εκπρόσωπο του αρμόδιου Υπουργείου της Σουηδικής Προεδρίας. Πρόκειται, θυμίζω, για μια διαδικασία συναπόφασης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν μπορεί να κλείσει τα συμπεράσματά του πριν ολοκληρώσουμε εμείς την πρώτη ανάγνωση. och ehm, jag lämnar ordet θα ήθελα να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην κυρία Εστρέλα για να μας παρουσιάσει το θέμα της. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να, ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την αλλαγή που κάναμε στη συζήτηση των σημείων της ημερήσιας διάταξης, ώστε να μετατοπίσουμε λίγο επί το νωρίτερο αυτό το θέμα για να προλάβω κι εγώ να επιστρέψω στη Λισαβόνα για να συμμετέχω στην πανηγυρική εκδήλωση που θα γίνει με την για την έναρξη της ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τους σκιώδεις ηγητές που συνέβαλα με τις προτάσεις τους και με την κριτική τους γνώμη στη διαμόρφωση της πρότασης ε, που καταθέτω στην έκθεσή μου. Τους τελευταίους μήνες συμμετείχα σε πολλές και διάφορες ε, συνεδριάσεις και διαβουλεύσεις με τους σκιώδεις ηγητές όπως ήταν προφανές πρώτα απ' όλα αλλά ταυτόχρονα και με εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με εκπροσώπους των συνδικάτων και οργανώσεων προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών. Δηλαδή, προσπάθησα να ακούσω όλους τους ενδιαφερόμενους ένα ευρύτατο φάσμα απόψεων για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας και ζήτησα από όλους ε, τις προτάσεις και τη συνεισφορά τους. Από όλες τις πολιτικές ομάδες έλαβα προτάσεις με εξαίρεση το ΕΛΚ. Τις προτάσεις αυτές τις ενσωμάτωσα ε, στην έκθεσή μου που σας υποβάλλω σήμερα και θα τη συζητήσουμε. Πρόθεσή μου ήταν να εξασφαλίσω όσο το δυνατό πιο ευρία συνένεση γίνεται Μία συνένεση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των γυναικών, των οικογενειών, στα συμφέροντα των παιδιών, αλλά και στις ανάγκες της κοινωνίας μας. Είναι αλήθεια ότι διανύουμε χαλεπούς αρούς, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι δεν νομοθετούμε πρόθεσμα για το παρόν και για το εγγύς μέλλον, αλλά νομοθετούμε για τις επόμενες δεκαετίες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η οδηγία έχει ήδη ηλικία 17 ετών. Δηλαδή, η νομοθεσία που θα θεσπίσουμε αναθεωρώντας την οδηγία αυτή θα διαρκέσει για πολλά χρόνια. Δεν γνωρίζουμε πόσα ακριβώς, αλλά σίγουρα μία δεκαετία τουλάχιστον, για να μην πω περισσότερες. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε κοντόφθαλμα, αλλά θα πρέπει να έχουμε ε, υπόψη μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Οι πιο σημαντικές προτάσεις της έκθεσής μου είναι γνωστές. Είναι 73 όλες οι προτάσεις. Οι πιο σημαντικές όμως σχετίζονται με την παράταση της άδειας μητρότητας. από τις 14 στις 20 εβδομάδες προτείνω εγώ. Τώρα προς το σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι μετά από διαβουλεύσεις και επαφές με πολλούς συναδέλφους και με εκπροσώπους των διαφόρων οργανώσεων που σας προανέφερα δήλωσα ότι είμαι πρόθυμη και διαλλακτική και αν αυτή είναι η δεδηλωμένη άποψη της πλειοψηφίας. Είμαι διατεθειμένη να κάνω μια περικοπή αυτής της πρότασής μου, ώστε ένα τμήμα να το διεκδικεί η γυναίκα και ένα τμήμα ο σύζυγος, οι άνδρες. Για παράδειγμα, συνάδελφοι, κάποιοι συνάδελφοι πρότειναν να προβλέψουμε 18 μήνες άδεια 18 ε, συγγνώμη, εβδομάδες άδεια μητρότητας και ή δύο επόμενες εβδομάδες μέχρι τις 20 να λαμβάνεται από το σύζυγο. Άλλοι πρότειναν 16 εβδομάδες να είναι η άδεια μητρότητας και να μπορεί να παραταθεί μέχρι 20 αρκεί οι δύο από αυτές τις εβδομάδες ε, να ληφθούν από το σύζυγο. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να εφαρμόσουμε στην οδηγία αυτή κάτι που ήδη ισχύει ως πρακτική σε ορισμένα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία. Στις χώρες αυτές ήδη υπάρχει αυτός ο καταμερισμός στην άδεια. Και το ζευγάρι μπορεί να αποφασίσει ποιος θα λάβει την άδεια και τη διάρκεια θα έχει αυτή ώστε με μεγαλύτερη ελευθερία και ελαστικότητα να μπορούν οι δύο σύζυγοι με κοινή συμφωνία να βρουν την καλύτερη λύση που θα τους εξυπηρετεί καλύτερα. Βέβαια, στόχος μας είναι ένας πιο δίκαιος καταμερισμός των οικογενειακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ώστε να υλοποιήσουμε το στόχο μας που είναι ο συνδυασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και για τους άνδρες αλλά και για τις γυναίκες. Πολύ πρόσφατα, γι' αυτό και δεν ε, κατάφερα να διαβάσω προσεκτικά όλη την έκθεση, έμαθα ότι το Σουηδικό Ινστιτούτο Έρευνας για την ε, Βιομηχανική Οικονομία εκπώνησε μια σχετική μελέτη ε, επισημένοντας ότι υπάρχουν λίγες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις ε, στο κράτος πρόνοιας και μάλιστα επισημαίνει η μελέτη ότι όσο πιο παρατεταμένη είναι η άδεια μητρότητας τόσο πιο ε, μικρές είναι οι πιθανότητες να φτάσει μια γυναίκα στο απόγειο της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας. Φαίνεται δηλαδή ότι η μητρότητα είναι ένα εμπόδιο στην επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών. Και φυσικά αυτό το θέμα δεν περιορίζεται μόνο στην άδεια μητρότητας, γιατί αυτή η άδεια περισσότερο στόχο έχει την αποκατάσταση της ισότητας ανδρών και γυναικών. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να προωθήσουμε και κάποιες κοινωνικές υποδομές όπως βρεφονιπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, σταθμούς φύλαξης παιδιών, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να εκπληρώσουν και τους επαγγελματικούς τους στόχους χωρίς αίσθημα ενοχής. Γιατί είναι απαράδεκτο να αναγκάζονται οι γυναίκες να διαλέξουν μεταξύ της μητρότητας και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Θα πρέπει να υπάρχουν συνθήκες για να μπορέσουν οι γυναίκες να συνδυάζουν αυτές τις πτυχές ε, της ζωής τους που είναι και οι πολύ σημαντικές και να εξορροπούν την επαγγελματική σταδιοδρομή και τον επαγγελματικό βίο με την ιδιωτική σφαίρα και την οικογενειακή ζωή. Επίσης είναι πολύ σημαντικό η γυναίκα στην άδεια μητρότητας τουλάχιστον στις πρώτες έξι εβδομάδες μετά το τοκετό να λαμβάνει ατόφια την αμοιβή της, να λαμβάνει πλήρη το μισθό γιατί αυτές οι πρώτες έξι εβδομάδες ε, κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την ε, αποκατάσταση της ε, υγείας της γυναίκας και την ανάνυψή της μετά τον τοκετό. Επίσης θα πρέπει να κατοχυρωθεί η αρχή της ε, πλήρους καταβολής του μισθού για τις πρώτες έξι εβδομάδες. Στις περιπτώσεις όμως που δεν θα είναι δυνατό κάτι τέτοιο, να εξασφαλιστεί τουλάχιστον η καταβολή του 80% του μισθού κατά τις έξι πρώτες εβδομάδες. Γιατί δεν θα πρέπει να πλήττονται οικονομικά οικογένειες επειδή κάνουν την επιλογή να αποκτήσουν παιδιά. Είναι στοιχειώδες θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης κάτι τέτοιο. Άλλωστε αντιβαίνει στον ευρωπαϊκό στόχο της παροχής κινήτρων για τη γεννητικότητα, αν πλήττονται οικονομικά οικογένειες που διαλέγουν να τεκνοποιήσουν. Άλλο θέμα είναι η κατοχήρωση της ε, επικουρικής άδειας μητρότητας ε, για, εξαιρετικές, για ιδιαίτερες περιστάσεις, εκεί που χρειάζεται δηλαδή περισσότερος ε, καιρός για την αποκατάσταση της υγείας, την ανάνυψη της γυναίκας μετά τον τοκετό. Επίσης, η συμπερίληψη των οικιακών βοηθών στο σύστημα που δεν έτυχαν προστασία. δεν είχαν καν δικαιώματα στον τομέα αυτό. Επίσης, απαγορεύεται η απόλυση μιας γυναίκας από την έναρξη της ε, εγκυμοσύνης μέχρι δύο μήνες μετά το τέλος ε, της λήξης της άδειας μητρότητας. Επίσης, η απαγόρευση της υποχρέωσης ε, υπερορι... άσκηση υπερορίας ή νυχτερινής εργασίας ανάγκη προστασίας της μητρότητας και σε περίπτωση υιοθεσία. Δηλαδή, οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και στην περίπτωση υιοθεσία. Προτείνω και μία προληπτική προσέγγιση της ε, αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της αναπαραγωγικής υγείας. Επιπλέον, προβλέπω το δικαίωμα στον ε, ημερήσιο χρόνο για το θυλασμό με βάση τις συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προτείνει να δώσουμε ενάυσματα για το θυλασμό. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτή η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας συνδυάζει ως νομική βάση το άρθρο 176 με το 141. Το πρώτο άρθρο αναφέρεται στα θέματα υγείας και το δεύτερο στα θέματα ισότητας. Δηλαδή, το πεδίο εφαρμογή οδηγία διευρύνθηκε με την αναθεώρηση αυτή, με το συνδυασμό των δύο νομικών βάσεων και έτσι μπορούμε να συντάξουμε κάποιες τροπολογίες που διευκολύνουν το συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή και την ιδιωτική ζωή. Πρόθεσή μου είναι να αναδείξουμε ένα νέο μοντέλο εργαζόμενων γονιών για να καταπολεμήσουμε το στερεότυπο που θέλει τη γυναίκα να είναι περισσότερο στο σπίτι και να τεκνοποιεί παρά ε, παρούσα στην αγορά εργασίας και να παραγάγει. Η γυναίκα δεν είναι μόνο μητέρα, είναι και εργαζόμενη. Δίνει το παρόν λοιπόν στην αγορά εργασίας και έχει αντίστοιχα δικαιώματα με τον άνδρα στην επαγγελματική αυτοεκπλήρωση. Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους ολοκληρώνοντας να συνεργαστούμε για να βρούμε από κοινού τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των οικογενειών, τις ανάγκες των παιδιών και της κοινωνίας, έχοντας φυσικά υπόψη ότι η αναθεώρηση της οδηγίας δεν έχει ως μοναδικό στόχο την προστασία των εγγύων λεχόνων ή γαλουχουσών γυναικών, αλλά έχει και μία άλλη πτυχή, την πτυχή της ε, προαγωγής της ισότητας των δύο φύλων. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Στρέλα. Ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Υπάρχει ήδη εδώ ένας κατάλογος εγγεγραμμένων ομιλητών, ομιλητριών. Η κυρία Λούλιν ξεκινάει. Καταρχά θα έπρεπε να πάρει πρώτη το λόγο νομίζω η κυρία Ζαμπόρσκα, η οποία είναι η σκιώδη εισηγήτρια, έτσι νομίζω. Έχετε δίκιο κυρία Ζαμπόσκα. Πρέπει να ομολογήσω ότι εγώ ε, δεν υπολόγισα ότι θα ασχοληθούμε με την έκθεση αυτή τόσο νωρίς το πρωί. Ε, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν ε, διαπιστώνω ότι πρόκειται εδώ για μία ένα νέο σχέδιο της ε, έκθεσης. Εγώ ε, είχα υπόψη μου την παλιά έκθεση και διαπιστώνω ότι κατ' ουσίαν εδώ πρόκειται για δύο ταυτόσιμα κείμενα. Δηλαδή οι αλλαγές είναι τόσο απειροελάχιστες που η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι αναγκασμένη να καταλήξει στο ότι η συγγήτρια δεν βελτίωσε το κείμενό της. Και λυπάμαι πάρα πολύ που η κυρία Εστρέλα δεν ε, δέχθηκε τα σχόλιά μας, τα οποία αναφέρθηκαν επανειλημμένα στις συζητήσεις μας. Στην έκθεση λοιπόν υπάρχουν ε, τρεις ε, μορφές άδειας η γονική, η μητρότητα. Ε, όλα αυτά, κατά την άποψή μου, οδηγούν σε χάος αυτές οι τρεις άδειε που αναφέρονται. Η κυρία Στρέρα αναφέρεται στην ισότητα των δύο φίλων, αλλά εδώ στην έκθεση που μας παρουσίασε, δυστυχώς, εκεί γίνεται λόγος μόνο για την άδεια μητρότητας. Ε, πρόκειται για την ε, προστασία των μητέρων ε, μετά τον τοκετό και κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν συμφωνήσει όσον αφορά τη γονεϊκή άδεια και αυτή τη στιγμή τρέχουν συζητήσεις των κοινωνικών εταίρων που αφορούν στην περίφημη οικογενειακή άδεια, όπως τη χαρακτηρίζουν, family leave εγώ εξ όσων γνωρίζω θα υποβληθεί και μια σχετική έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία εισηγήτρια είπε ότι κατά την προετοιμασία της έκθεσης ε, διεξήγαγε συζητήσεις με το Συμβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με διάφορους οργανισμούς και η δική μας η πολιτική ομάδα συζήτησε με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς είχαμε συζητήσεις με εκπροσώπους οργανισμών γυναικών και της οικογένειας. Και τελικά καταλήξαμε στο ότι είναι απαραίτητο στην έκθεση αυτή να μην γίνεται μπέρδεμα με τις τρεις μορφές άδειας, να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κατόπιν τούτου πρότεινα αυτό βέβαια που είπε η συγγήτρια ότι ε, πρέπει να έχουμε ένα σύγχρονο κείμενο. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες, θέλουμε το θέμα της μητρότητας ε, να το εξετάσουμε με έναν τρόπο πιο σύγχρονο, με το ε, βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ. Η έκθεση που μας έχει κατατεθεί δεν ε, μας ικανοποιεί. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω η Επιτροπή μας να συζητήσει για την έκθεση αυτή όταν θα έχουμε μπροστά μας το κείμενο και των τριών οδηγιών, δηλαδή οδηγία για τη μητρότητα για την άδεια μητρότητας, για την άδεια οικογένειας και για την άδεια πατρότητας και νομίζω ότι τότε θα μπορούμε να συζητήσουμε και να αναζητήσουμε συγκεκριμένες λύσεις. Πραγματικά θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν τελικά δεν θα ήθελε που δεν η Ολομέλεια να απορρίψει για άλλη μια φορά αυτή την έκθεση. Αυτό δεν θα το ήθελε που δεν Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ζεμπόσκα. Περνώ τώρα στον κανονικό κατάλογο μιλητών και δίνω το λόγο στην κυρία Λούκας. Μετά θα μιλήσω κι εγώ και η κυρία Μποσκούρτ. Λούκας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μειοψηφία. Θα στηρίξω λοιπόν την πρόταση της κυρία Εστρέλα. Νομίζω ότι το θέμα είναι να βρούμε ποια είναι η πλειοψηφία σε αυτό το κοινοβούλιο. Αυτό κάνει η κυρία Στρέλα και νομίζω ότι έχει δίκιο ότι τα στοιχεία τα οποία στέλνει μέσω της έκθεσής της στην Ολομέλεια είναι τα σωστά. Σχετικά με την διεύρυνση της εμβέλειας, αν θέλετε, αυτής της οδηγίας και της νομικής της βάσης, αυτό είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί το Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συζητά θέματα όπως τον εξυγχρονισμό της γονεϊκής άδεια και νομίζω ότι ο μοναδικός τρόπος του εξυγχρονισμού αυτού είναι να το προσαρμόσει στον τρόπο ζωής του κόσμου σήμερα. Ακριβώς αυτό που κάνει η κυρία Εστρέλα. Εγώ και η ομάδα μου λοιπόν υποστηρίζουμε αυτήν την υποχρεωτικά πληρωμένη ε, εναλλακτική άδεια δύο εβδομάδων και πρέπει να είναι η πληρωμή υποχρεωτική γιατί αλλιώς ε, δεν θα την επιλέγει ο κόσμος. Το θέμα δεν είναι να εμένουμε σε αφηρημένες ιδανικές καταστάσεις όπως καλύτερες συνθήκες κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να διευκολύνουμε με συγκεκριμένο τρόπο την διευκόλυνση των ε, ε, μητέρων και των γονιών γενικότερα. Μόνο έτσι θα επιδιώξουμε να γίνουν οι πολιτικές της Ένωσης προοδευτικές. Αυτό κάνει η πρόταση Εστρέλα, παίρνει συγκεκριμένα μέτρα, όχι θεωρητικά, νομικά μέτρα, πρακτικά που θα βοηθήσουν το κοινό. Σχετικά με το θυλασμό, αυτά τα οποία λέγονται τα βρίσκω πάρα πολύ θετικά. Εδώ και 15 χρόνια με έδιωξαν από ένα δημοτικό συμβούλιο γιατί εγώ θύλαζα το παιδί μου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και με έδιωξαν από την αίθουσα. Καταλαβαίνετε τι οδυνηρή διαδικασία ήταν αυτή την οποία έζησα. Μια αλλαγή την οποία θα θέλαμε, όπως γνωρίζει η κυρία Εστρέλα, είναι η διάρκεια της άδεια. Οι 18 εβδομάδες είναι δεδομένο για τις περισσότερες χώρες και μία αύξηση από τις 14 στις 18 στους 18 μήνες για ορισμένες χώρες δεν είναι κάτι το σημαντικό. Σε πολλές χώρες έχουμε πολύ μεγαλύτερε φιλοδοξίες θα έλεγα και γι' αυτό θα ήθελα να γίνει δεκτή η τροπολογία μας η οποία στοχεύει τις 24 εβδομάδες. Νομίζουμε ότι ο στόχος των 24 εβδομάδων είναι ορθότερος. Τελειώνοντας, Ελπίζω να συνεργαστούμε σωστά με τους συναδέλφους στην Επιτροπή Απασχόλησης και θα ήθελα να ζητήσω από τις πολιτικές ομάδες να συνεργάζονται με τους ομολόγους τους στην Επιτροπή Απασχόλησης έτσι ώστε να περάσει από την Ολομέλεια γιατί πολλοί είναι ο κόσμος ο οποίος προσδοκά να γίνουν πραγματικότητα αυτά που προτείνουμε. Σας ευχαριστώ κυρία Λούκας. είχα και εγώ δώσει το όνομά μου. Κάποιες παρατηρήσεις πρώτες θα ήθελα να κάνω και να θέσω και κάποιες ερωτήσεις. Στο κείμενο ε, αναφέρεστε σε υποχρεωτική άδεια. Διαρωτώ με εδώ. Ίσως αντί να γράψουμε τη λέξη υποχρεωτική, μήπως να μιλήσουμε για δικαίωμα δικαίωμα σε άδεια. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο να το κάνουμε έτσι, να διευκρινίσουμε ότι μπορεί να αφορά τη μητέρα ή τον πατέρα, αλλά είναι ένα δικαίωμα περισσότερο ε, του ε, εργαζομένου ή της εργαζομένης. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο όρος υποχρεωτική ε, δεν είναι σωστό. Η άδεια είναι ένα δικαίωμα και δικαιούται κανείς να πάρει την άδεια αυτή η οποία του αναλογεί. Ένα δικαίωμα το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται με ισότιμο τρόπο και στις γυναίκες και στους άνδρες. Καταλαβαίνω βέβαια ότι πίσω από το επίθετο υποχρεωτικός, υποχρεωτική, εσείς έχετε σαν στόχο την προστασία των εργαζομένων, για να το πω καλύτερα, την προστασία του ιδίου του δικαιώματος το οποίο έχουν. Παρ' όλα αυτά ε, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ο εργαζόμενος και οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα που έχουν σε μία συγκεκριμένη άδεια. Άλλο σημείο. Οι έξι εβδομάδες υποχρεωτικής. Πάλι εδώ έρχεται ο όρος υποχρεωτική άδεια. Εφόσον εμένουμε στο συγκεκριμένο επίθετο, αυτό ε, λέγει ότι μόνον η μητέρα μπορεί να πάρει τις έξι αυτές εβδομάδες. Ενώ έχουμε επανειλημμένα πει στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής ότι αυτό πρέπει να αφορά ε, και τα δύο φύλλα. Και νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ε, ισότητας. Η ευθύνη δηλαδή του παιδιού ε, δεν είναι αποκλειστικότητα της μητέρας αλλά και του πατέρα. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για υποχρεωτική άδεια της μητέρας. Αλλά είναι ένα δικαίωμα για την γυναίκα ή τον άνδρα, για τη μητέρα ή τον πατέρα. Έχουμε μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι στις χώρες τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα την άδεια αυτή να πάρει ο πατέρας του παιδιού, αυτό επηρεάζει θετικά την ισότητα ανδρών γυναικών. Στο μέλλον, μιας και γνωρίζουμε την μεγάλη σημασία που έχει το να είναι ισότιμα συμμέτοχοι στην κοινωνική ζωή και στον επαγγελματικό κόσμο οι άνδρες και οι γυναίκες, διαπιστώνουμε δυστυχώς σήμερα και ότι πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες εργάζονται φέρουν τεράστιες ε, ευθύνες γύρω από την οικογενειακή ζωή, γύρω από τις οικογενειακές ευθύνες, γύρω από αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς μη αμοιβόμενη ουσιαστικά εργασία. Ενώ αν δίνουμε τη δυνατότητα εξ αρχής στους πατέρες ε, να αναλαμβάνουν τις οικογενειακές τους ευθύνες εκ των προτέρων επαναλαμβάνω, τότε θα υπάρξει μια σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων και στον τομέα αυτής της μη αμοιβόμενης εργασίας όπως η φροντίδα των παιδιών και η ουσιαστική συμμετοχή στην οικογενειακή δραστηριότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ευκταίο και απαραίτητο θα έλεγα όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και τους γονείς είναι κάτι το οποίο πλουτίζει την ζωή μας είναι κάτι το οποίο επιτρέπει να υπάρχει μια ικανοποιητική κοινωνική ζωή και μια ικανοποιητική οικογενειακή ε, ζωή τώρα για τον θυλασμό. Κατανοώ και συμμερίζομαι εν πολύ στην άποψη της κυρίας Λούκας οι γυναίκες οι οποίες επιλέγουν τον θυλασμό θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν και την διάρκεια του. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα για τις ε, θυλάζουσες γυναίκες να φέρουν εις πέρα στη συγκεκριμένη αυτή επιλογή τους. Θυμίζω ότι ήδη από το 2002 ο ε, ε, Διεθνής Οργανισμός Υγείας έχει υπογραμμίσει ότι ο θυλασμός ε, είναι η καλύτερη λύση για την ανατροφή των παιδιών, των μικρών παιδιών και θα πρέπει να διαρκεί έξι μήνες τουλάχιστον. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν το θέμα αυτό και αυτό φαίνεται από τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας και προφανώς αυτές οι συστάσεις είναι καρπός μια συζήτηση η οποία έχει γίνει. Υπάρχουν, ξέρετε, διάφορα προϊόντα υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος και σε πολλές χώρες κυκλοφορούν διάφορα γάλατα τα οποία ονομάζονται α, ακριβώς μητρικού τύπου θα έλεγα ενώ σε καμία περίπτωση δεν προσφέρουν στο παιδί ε, τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία τα οποία του είναι απαραίτητα για την ανατροφή του. Συνεπώς, η σύσταση αυτή του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας αφορά κυρίως τα παιδιά στις ε, ε, υποανάπτυξη χώρες, περισσότερο από κάτι άλλο και δεν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καθιστούμε ε, θύματα ή ένοχες, να τις κάνουμε να νιώθουν ένοχες τις γυναίκες οι οποίες δεν επιλέγουν ή δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι κάτι το επιθυμητό εφόσον οι γυναίκες το επιθυμούν και δίνανται να θυλάσουν. Αλλά δεν θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να θυλάζουμε μέχρι έξι μήνες. Θα πρέπει η επιλογή να γίνεται από τις ίδιες τις μητέρες. Και θυμίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να φυλάζουν για έξι μήνες. Δεν θα πρέπει λοιπόν σε μια πρόταση οδηγίας να δώσουμε την εικόνα ότι στις γυναίκες αυτές οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα του θυλασμού δεν είναι γυναίκες που φροντίζουν σωστά τα παιδιά τους, που μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά τους. Και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε να εννοηθεί ότι τα παιδιά έχουν μικρότερες δυνατότητες όταν δεν είναι σε θέση να θυλάσουν. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια διαφορετική λύση για την λέξη υποχρεωτικός και να μιλήσουμε για δικαίωμα. Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Μπόσκουρθ και μετά η κυρία Λούλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ε, υπενθυμίσω ότι η έκθεση αυτή δεν απορρίφθηκε στην Ολομέλεια, δεν είναι αλήθεια αυτό, απλά αναβλήθηκε, μετατέθηκε και η ψηφοφορία εκρεμεί. Εγώ λοιπόν θα ήθελα έτσι κι αλλιώς να ευχαριστήσω την ε, κυρία Στρέλα, την εισηγήτριά μας, για το γεγονός ότι συμφώνησε με όλες τις πολιτικές ομάδες για να βελτιώσει την έκθεση. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η έκθεση έχει βελτιωθεί και τώρα αποτελεί πραγματικό εργαλείο εργασίας. Πρόκειται για την πρόσπιση των συμφερόντων των ε, γυναικών, ε, των μητέρων. Πράγματι, στην έκθεση αυτή ε, δεν γίνεται λόγος μόνο για τη μητέρα, γίνεται λόγος και για τον πατέρα και για τον σύντροφο δεν πρόκειται μόνο για τη μητέρα. Πάμε πολύ, αλλά ο κόσμος δεν αποτελείται μόνο από μητέρες, υπάρχουν και άλλα ανθρώπινα όντα. Και συμφωνώ με την κυρία Σβένσεν με αυτό που είπε, ε, που τοποθετήθηκε επί του ε, επιθέτου υποχρεωτικός. Και εγώ ε, πιστεύω ότι ήταν καλύτερα να μην μιλάμε για υποχρέωση, αλλά να μιλάμε για δικαίωμα, το οποίο μπορεί κανείς να διεκδικήσει. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι μια πολύ καλή τροποποίηση. Εγώ αυτά είχα να σας πω και κατά τα άλλα ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και να εγκρίνουμε τελικά αυτήν την έκθεση. Πρόκειται για τα συμφέροντα πάρα πολλών ανθρώπων, συμφέροντα πατέρων, μητέρων, ε, συντρόφων και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε όλα αυτά κατά νου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. κυρία Μπόσκουτ, η κυρία Λούλινγκ έχει τώρα το λόγο και μετά η κυρία Κλάς. Η κυρία Λούλινγκ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω εδώ ότι η οδηγία έχει στόχο την ε, βελτίωση της ε, υγείας και της ασφάλειας των εγγύων, λεχόνων και γαλουχουσών γυναικών στο χώρο εργασίας τους. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα δεύτερο σχέδιο έκθεση, αλλά για ένα σχέδιο έκθεσης, γιατί έκθεση θα είναι, δεν θα είναι δεύτερη έκθεση. Γιατί η πρώτη αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή. Η κυρία Στρέλα έχει ένα σπάνιο ταλέντο υπερφόρτωσης της έκθεσής της με σχόλια που είναι τελείως άσχετα με το θέμα της οδηγίας και εκτός τόπου και χρόνου τελείως ακατάλληλα για ένα νομοθετικό κείμενο. Δεν έχουμε εδώ ένα κατάλογο αγορών, ένα shopping list. Δεν είναι αυτό το περιεχόμενο της έκθεσης. Θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα νομοθετικό κείμενο που θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Και είναι αδύνατο με τέτοιες προτάσεις να φτάσουμε σε ένα σωστό νομοθετικό κείμενο. Δεν ε, κατέθεσα τροπολογίες από βίτσιο, γιατί αν σκεφτείτε πώς, τι κόστος θα έχουν αυτές οι ασυνάρτητες παράλογες και ανεφάρμοστες, ανέφικτες ε, προτάσεις, τι να σας πω. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία ιδέα ούτε για το εργατικό δίκαιο, ούτε για τις συλλογικέ ε, διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για ένα συνοθήλευμα προτάσεων που μια έκθεση, πρόκειται για μια έκθεση που βρήθη επαναλήψεων και αντιφάσεων και εγώ θα πρότεινα νέα αναπομπή της έκθεσης, προκειμένου να επικεντρωθούμε στο γνήσιο στόχο της πρότασης οδηγίας. Γιατί έχουμε απομακρυνθεί από αυτόν. Έχω την αίσθηση ακούγοντας τις παρατηρήσεις ε, των μελών της Επιτροπής και ακούγοντας ιδιαίτερα εσάς κυρία Πρόεδρε ότι ζούμε σε τελείως διαφορετικό κόσμο. Γιατί <laughs> από ό,τι ξέρω, οι γυναίκες εγκυμονούν και όχι οι άνδρες, εκτός πια και αν έρθουν τα πάνω κάτω. Οι γυναίκες φέρουν στον κόσμο τα παιδιά. Διαβάζοντας τις προτάσεις σας, βλέπω ότι το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσετε το δικαίωμα αναπαραγωγή των ανδρών και τα δικαιώματα άδεια πατρότητα. Νομίζω ότι αυτό σα ενδιαφέρει περισσότερο από την προστασία τη μητρότητα. Τέτοιου είδου θεωρίε είναι ιδιαίτερα επικίνδυνε και ιδιαίτερα η θεωρία σα ότι δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική άδεια, αυτή και αν είναι επικίνδυνη. Δώσαμε μάχη για δεκαετίες ολόκληρες. Εγώ συνέταξα την πρώτη έκθεση για την προστασία της μητρότητας το 1966. Δώσαμε μάχη για να κατοχυρώσουμε υποχρεωτικά την άδεια μητρότητας, για να προστατεύσουμε την υγεία της μητέρας και του παιδιού πριν και μετά τον τοκετό. Και τώρα θέλετε όλα αυτά να τα ανατρέψετε, να τα διαλύσετε. Θα πρέπει να το καλοσκεφτείτε νομίζω. Πραγματικά θα πρέπει να ξεδιαλύνετε τους στόχους σας πρώτα απ' όλα και να αντιληφθείτε τον κίνδυνο που δημιουργείται για την προστασία των γυναικών και των παιδιών. Θα σου ομολογώ ότι για μένα το κείμενο είναι ανέφικτο και ζητώ αναπομπή και τροποποίηση της έκθεσης Άρδιν. Βέβαια, μας λέτε ότι είμαστε μειοψηφία, αλλά θα τα δούμε. Πάντως, αν η πλειοψηφία της Επιτροπής ε, Γυναικών θέλει να εγκρίνει αυτή την ασυναρτησία, τι να σας πω. Καλή τύχη σας εύχομαι για τη συνδιαλλαγή, αν καταφέρετε να φτάσετε μέχρι εκεί. Πάντως, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να παρεμποδίσω την πρόωθηση μιας τέτοιας πρότασης. Δεν θα ήθελα να υποβληθεί αυτή η πρόταση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Γιατί θα γελιοποιήσει την Επιτροπή Γυναικών μια τέτοια πρόταση. Ούτω ή άλλω δεν μα παίρνουν στα σοβαρά, αλλά με τέτοιου είδου εκθέσει τότε είναι που θα γίνουμε ρεντίκολο και στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί λοιπόν να μην επικεντρωθούμε στο θέμα τη προστασίας της μητρότητας γιατί οι κοινωνικοί εταίροι έχουν διαπραγματεύσεις για την άδεια πατρότητας. Οι κοινωνικοί εταίροι ήδη είχαν διαπραγματεύσεις για τη γονική άδεια. Και μάλιστα έχουμε λάβει το κείμενο και έχουμε συντάξει και ψήφισμα. Θα βελτιωθεί η νομοθεσία μας για την άδεια πατρότητας, ούτως ή άλλως. Γιατί θέλετε σώνει και καλά στο δικό σας κείμενο να κάνετε ένα τέτοιο ανακάτεμα που θα είναι τόσο δύσχριστο και ανέφικτο στην πράξη. Γι' αυτό λέω αναπομπή, ρηξικέλευτη τροποποίηση της έκθεσης και επικέντρωση στα ουσιώδη. Γιατί αν πραγματικά θέλετε να καθυστερήσετε την προτινόμενη μεταρρύθμιση, τότε είναι που πρέπει να συντάσσετε τις εκθέσεις τη δική σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λούλινγκ. Η κυρία Κλάς έχει το λόγο και μετά η κυρία Καρθία Κουτιέρες. Κυρία Κλάς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Ζαμπόφσκα. Τελικά τι γίνεται εδώ, στρεφόμαστε γύρω από ένα πράγμα, γυρίζουμε γύρω-γύρω από αυτό και τίποτα δεν βελτιώνεται. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συζητήσουμε για την ουσία. Κοιτάξτε, η Επιτροπή έχει νέα σύσταση και τώρα λοιπόν απευθύνομαι στα νέα μέλη που είναι για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ λοιπόν να σκεφτούν τα θεμελιώδη θέματα. Δηλαδή, Κατά την άποψή μας, πού είναι απαραίτητο να υπάρχει ισότητα των δύο φύλων. Η κυρία Λούλινγκ το είπε πάρα πολύ καλά. Καλύτερα δεν γίνεται. Και εγώ συμμερίζομαι αυτό το φόβο, το φόβο ότι ως γυναίκες εκχωρούμε κάτι το οποίο ούτε καν μπορούμε να εκχωρήσουμε. Μα είναι το μοναδικό δικαίωμα το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο εμάς τις γυναίκες. Εμείς είμαστε τα ανθρώπινα κοινά όντα που χαρίζουν τη ζωή, που το φέρνουν στον κόσμο. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το μοιραστεί και αυτή η οδηγία αφορά τη βελτίωση και την ασφάλεια, την προστασία υγείας των εργαζομένων γυναικών, των γαλουχουσών ε, στο χώρο εργασίας. Σωστά λοιπόν αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο η οδηγία και η τροπολογία και εμείς τι θα κάνουμε, θα την αποδυναμώσουμε με το να συμπεριλάβουμε και άνδρες. Μα δεν γίνεται αυτό. Ούτε η φύση έχει προβλέψει γι' αυτό. Είναι αφύσικο, δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ θερμά να διατηρήσουμε αυτό το δικαίωμα το οποίο διεκδίκησαν με αγώνες οι προκάτοχοί μας σε αυτήν την Επιτροπή. Και το πετύχαμε και μετά θα πρέπει να δούμε πώς αυτό το δικαίωμα μπορούμε να το διατηρήσουμε στις ε, σημερινές συνθήκες, να το διακοσμήσουμε, να το επεκτείνουμε. Γιατί στη συζήτηση έχουν τεθεί και άλλα θέματα. Δηλαδή, έχει τεθεί το έχεις ερώτημα, μα είναι αρμόδια η Ευρώπη για αυτό το θέμα. Ας το σκεφτούμε λιγάκι. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διαφορετικά ε, κοινωνικά συστήματα ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που είναι ανοιχτά. Α δούμε το Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο, παραδείγματο χάρη, η ε, προστασία τη ε, μητρότητα ε, πλημμυρίζεται από φορολογικέ ρυθμίσει και καλύπτεται όμω από του φόρου. Σε εμά, στη Γερμανία, οι εργοδότε είναι εκείνοι που πληρώνουν για την άδεια μητρότητα. Μιλάμε για ένα ποσό περίπου των 700 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα συμπεριλάβουμε. Δηλαδή, εμείς τελικά τι κινδυνεύουμε να κάνουμε. Πάμε να οικοδομήσουμε πάνω σε σαφρά θεμέλια, πάνω σε κάτι που δεν υφίσταται. Δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί η νομική βάση. Ω εκ τούτου, το πρώτο που θέλω να πω, αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε επιτύχει, να βασιστούμε στην παλιά οδηγία και αυτό να το κάνουμε πολύ προσεκτικά. Σήμερα ερωτάζουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας που μας αποδίδει περισσότερα δικαιώματα στο Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου είχαμε δικαιώματα, θα λάβουμε και άλλα. Πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε υπευθυνότητα για τις γυναίκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό κάνω έκκληση σε όλους αυτή τη στάση να κρατήσουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε κύριε Κλάς. Το λόγο έχει η κυρία Γκαρσία Πέρες και μετά η κυρία Βέρ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε όποια πολιτική παράταξη και αν ανήκει το κάθε μέλος της Επιτροπής, όλοι συμφωνούμε για την ευθύνη που φέρει η Επιτροπή μας για τη θέση εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας. Δεν συμφωνώ όμως να θεωρούμε ότι ο καθένας είναι υπεύθυνο μόνο όταν υποστηρίζει μια συγκεκριμένη άποψη και όλοι οι υπόλοιποι είναι ανεύθυνοι. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να ακούσουμε και να σεβαστούμε και τις αντίθετες απόψεις. Μπορεί ο καθένας έχει τη γνώμη του. Δεν δέχομαι όμως κάποιος να κρίνει τη δική μου γνώμη επικίνδυνη ή όπως αλλιώς τη χαρακτηρίζει. Θα πρέπει να αποστασιοποιηθούμε κάπως και να σεβαστούμε και τις διαφορές. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, θα πρέπει να τις σεβαστούμε. Σίγουρα μιλάμε για μια οδηγία περιμετρότητας και όλα τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών θέλουν να υπερασπίσουν τη μητρότητα. Θέλουμε όμως οι γυναίκες να βρίσκονται σε ισότιμη θέση με τους άνδρες για να μπορούν και να διαδραματίσουν το ρόλο τους ως μητέρες αλλά να έχουν δικαίωμα πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και η κατοχήρωση της άδειας πατρότητας δίνει την ευκαιρία και στους άνδρες και στις γυναίκες ε, να είναι ισοδύναμοι σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας. Όταν μια νεαρή γυναίκα πηγαίνει στη συνέντευξη εργασίας και ζητήσει μια αγορά εργασίας, η πρώτη ερώτηση είναι αν είναι παντρεμένη ή ανήπαντρη. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν σκοπεύει να γίνει μητέρα σύντομα. Ενώ ένας νεαρός ε, άνδρας δεν πρόκειται να απαντήσει σε τέτοιες ερωτήσεις σε μια συνέντευξη εργασίας. Γιατί ο εργοδότης ε, ξέρει ότι δεν θα του λείψει ο εργαζόμενος του για άδεια πατρότητες, Δεν θα τον στερηθεί. Οπότε αν σημειώσουμε κάποια πρόοδο στο θέμα της άδειας πατρότητας ώστε να εξορροπηθούν οι ρόλοι μεταξύ ανδρών και γυναικών και θα συμφιλιώσουμε την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή και θα αποκαταστήσουμε μια ισορροπία μεταξύ του ζευγαριού, ώστε και οι δύο να έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν τα παιδιά και να μεριμνούν για αυτά στι πρώτε ημέρε και εβδομάδε τη ζωή του. Γιατί ο συνδυασμό αυτό επαγγελματική και οικογενειακή ζωή δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τι γυναίκε, αλλά και του άντρε. Σίγουρα οι γυναίκε είναι οι μητέρε, αλλά και οι μητέρε χρειάζονται σε αυτέ τι πρώτε μέρε ε, τη ζωή των παιδιών του ε, μια συμπαράσταση από το σύζυγο, από το σύντροφο να μπορούν να μοιράζονται μαζί του τις οικογενειακές ευθύνες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα αυτό και να συμπεριλάβουμε στην οδηγία και τη δυνατότητα άδειας πατρότητας. Τώρα, αν δεν θέλουμε να τη χαρακτηρίσουμε υποχρεωτική ή να πούμε μία άδεια πατρότητας μεταποδοχών. Στην περίπτωση της Ισπανίας είχαμε πριν από μερικά χρόνια τη δυνατότητα για τον άνδρα να αναλάβει ένα τμήμα της άδεια μητρότητας. Αλλά κανένας δεν διεκδικούσε αυτό το δικαίωμα, κανένας άνδρας δεν το ζήτησε. Όταν προτάθηκε όμως ε, μεταποδοχών άδεια πατρότητας, ήδη το πρώτο χρόνο εφαρμογής, το 80% των ανδρών που έγιναν πατέρες, εποφελήθηκαν από αυτή τη διάταξη για την άδεια πατρότητας. Ακριβώς επειδή ήταν μεταποδοχών. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη αυτό το στοιχείο. Σε ό,τι αφορά το θέμα της γαλουχίας. Αν καταφέρουμε στο κείμενο αυτό να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και να διευκολύνουμε κάποιες αλλαγές, γιατί να μην το κάνουμε. Τίποτα δεν είναι αποκρισταλωμένο. Μπορούμε να συζητήσουμε, να καταλήξουμε σε πιο συνενετικές απόψεις. Για το θέμα της γαλουχίας μπορεί να υπάρχει και άλλη δυνατότητα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιες εθνικές νομοθεσίες να προβλέπουν κάποια περίοδο γαλουχίας ή ε, ημερήσια πάυση για το θυλασμό οι γυναίκες που δεν μπορούν να θυλάσουν αυτές τις ώρες ε, που προβλέπονται στην για την πάυση του θυλασμού μπορούν να τις συσσωρεύουν. Από τη στιγμή που έχει λήξει η άδεια πατρότητας, για δύο μέρες, ε, για δύο μήνες, συγγνώμη, η γυναίκα δικαιούται μία ώρα ε, θυλασμού τη μέρα ή μπορεί να τη συγκεντρώσει στο τέλος και να συγκεντρώσει μία εβδομάδα για να παραμείνει επιπλέον στο σπίτι. Θα δούμε, θα δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε ώστε οι γυναίκες που δεν θυλάζουν να μπορέσουν να, να συγκεντρώσουν αυτές τις ε, ώρες θυλασμού. Θα ήθελα να σας ζητήσω κατανόηση γιατί εγώ έχω κατανόηση προς τις αντίθετες απόψεις προς τις διαφορετικές απόψεις. Μιλήσαμε για 24 εβδομάδες, άλλοι μίλησαν για 18, άλλοι μίλησαν για 20 εβδομάδες, για δύο εβδομάδες πατρότητας. Πιστεύω ότι μπορούμε να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε συμφωνία που είναι σημαντική και για την υγεία της μητέρας. Γιατί καλό θα είναι κάποιος που αποφάσισε να κάνει οικογένεια να μπορεί να μοιραστεί με τον σύντροφο τη μέρημνα των παιδιών και τις οικογενειακές ευθύνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκαρσία Πέρας. Ευχαριστούμε πολύ και επόμενη ε, η κυρία Οβή. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει με ορισμένα από αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ε, ομιλητές και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι Ζούμε στον 21ο αιώνα βεβαίως ε, και πρέπει να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε επιτύχει αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η οδηγία είναι πλέον απαρχαιωμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να την εξυγχρονίσουμε, να την βελτιώσουμε και τούτο κυρίως διότι οι σημερινές μας αποφάσεις ε, θα επηρεάσουν το μέλλον, το απότερο μέλλον, όχι απαραίτητα το εγγύς μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν αφορούν ένα πράγμα. Αφορούν στην προστασία της μητρότητας. Το θέμα αυτό το συζητήσαμε και στην ομάδα μας και όσον αφορά την ιδεολογία σχετικά με την ε, άδεια πατρότητα. Το θέμα δεν είναι μόνο να δώσουμε άδεια στον πατέρα, αλλά να προστατεύσουμε την υγεία της μητέρας σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το σύνολο της οικογένειας, όταν δηλαδή το παιδί είναι πολύ μικρό. Ίσως ε, θα πρέπει να συζητήσουμε το δικαίωμα των πατέρων να ε, παίρνουν άδεια μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ίσως πράγματι το κράτος ε, να αναλάβει την υποχρέωση ε, χορήγησης ε, αδειά σε δύο εβδομάδες στον πατέρα. Και αυτές τις δύο εβδομάδες να μπορεί ίσως η ίδια η οικογένεια να αποφασίζει πότε θα τις διεκδικεί ο πατέρας. Μερικές φορές η υγεία της μητέρας επιδεινώνεται όχι τις αμέσως δύο επόμενες εβδομάδες μετά τον τοκετό αλλά κάποια στιγμή αργότερα όπου αισθάνονται οι μητέρες ε, κουρασμένες, έχουν προβλήματα με το θυλασμό και εκεί ίσως χρειάζονται κάποια στήριξη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να συζητήσουμε είναι το δικαίωμα των πατέρων να έχουν αυτή την άδεια, την υποχρέωση του κράτους να καλύπτει αυτή την άδεια με αποδοχές, αλλά εγώ στηρίζω το θέμα της πατρότητας γιατί έχει άμεση σχέση με τη μητρότητα. Εξάλλου πρόκειται και για ένα θέμα ισότητας των δύο φύλων και δικαιοσύνης. Η προσέγγιση με την οποία αγνοούμε όλα αυτά και προσπαθούμε να καθυστερήσουμε το όλο θέμα, να επιλύσουμε το πρόβλημα μέσα από άλλες οδηγίες, αυτά όλα επιδεινώνουν την κατάσταση. Εκείνο λοιπόν που είναι απαραίτητο να υπάρχει είναι θέματα τα οποία έχουν ε, σχέση με το ίδιο θέμα. Και όταν πράγματα σχετίζονται μεταξύ του πρέπει να παρουσιάζονται και στο ίδιο έγγραφο. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ κυρία Οβίρ. Ε, θα δώσω το λόγο τώρα. Στην εισηγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης. Μετά η κυρία Κώστα, η κυρία Τόμψον και η κυρία Σαμπόσκα. Η εισηγήτρια όμως της Επιτροπής Απασχόλησης έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι εισηγήτρια της Συναρμόδιας Επιτροπής Απασχόλησης γύρω από το σχέδιο οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΝΤΙΤ Είχαμε πολύ στενή συνεργασία. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, τίθεται σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι και η εθνική γιορτή της Ρουμανίας. και όχι μόνο οι Ρουμάνες αλλά όλες οι Ευρωπαίες γυναίκες αξίζουν μια καλύτερη ζωή. Ιδιαίτερα για τις ε, νεότερες χώρες μέλη έχουμε ολοκληρώσει μια εικοσαετία μεταρρυθμίσεων, πολλές φορές οδυνηρών μεταρρυθμίσεων και καιρός είναι τώρα να υπάρξουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και στην ποιότητα της ζωής των γυναικών λέει η κυρία Πλάμπ από τη Ρωμανία. Το θέμα λοιπόν της ε, ισότητας ανδρών γυναικών δεν πρέπει να μείνει μια συζήτηση αλλά να γίνει μια πραγματικότητα. Η 1η λοιπόν Δεκεμβρίου του 2009 σημαίνει αυξημένες αρμοδιότητες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα των ανδρών και των γυναικών όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο και γι' αυτό ακριβώς υποστηρίζω την έκθεση την οποία προτείνει η Edit. Σημερίζομαι το όραμα της εισηγήτριας και τη στήριξα κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαμε στην Επιτροπή Απασχόλησης. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία είπαν και οι προηγούμενες συνάδελφοι. Είναι φυσικό να εκφράζονται διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις. Έχω την αίσθηση ότι έτσι και αλλιώς όλοι οι ευρωβουλευτές πρέπει να επιδεικνύουν την απαιτούμενη ευελιξία και να αναλαμβάνουν τις πολιτικές τους ευθύνες στα πλαίσια της συζήτησης ε, γύρω από την ποιότητα της ζωής των γυναικών στην Ευρώπη. Σε καμία περίπτωση αυτή η πρόταση δεν είναι ένας κατάλογος ευχών, είναι ένα ρεαλιστικό έγγραφο, είναι ένα έγγραφο το οποίο επιδέχεται φυσικά τροπολογήσεων. Φυσικά βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας της γυναίκας στο χώρο εργασίας. Και αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις γυναίκες οι οποίες είναι λεχόνες, τις γυναίκες οι οποίες είναι έγκυοι και τις γυναίκες που θυλάζουν. Ανησυχούμε όμως και με το θέμα της ισότιμης αντιμετώπισης ανδρών και γυναικών η νομική βάση είναι το άρθρο 141 και με βάση το συγκεκριμένο άρθρο θεωρώ ότι η πατρική άδεια θα πρέπει να συμπεριληφθεί ε, στην οδηγία αυτή αρκεί να επιδείξουμε την απαιτούμενη πολιτική βούληση. Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική βελτίωση, πρέπει να καταλήξουμε σε μια προοδευτικότερη Έκθεση. Συζητήσατε και για το αν η υποχρεωτική περίοδος της αδειοδότησης μετά τον τοκετό θα πρέπει να είναι έξι εβδομάδες ή όχι. Την προηγούμενη εβδομάδα να σας θυμίσω ότι το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή των συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η 183 σύσταση λέγει ότι η άδεια για τη μητέρα θα πρέπει να ληφθεί μέσα σε έξι εβδομάδες αμέσως μετά τον τοκετό. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την βασική αρχή των έξι εβδομάδων μετά τον τοκετό και σχετικά τώρα με την άδεια μητρότητα και με το επίδομα μητρότητας η Επιτροπή Απασχόλησης θεωρεί ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η πλήρης αμοιβή κατά τη διάρκεια του συνόλου της άδεια μητρότητας. Προφανώς και υπάρχουν διαφορετικές θέσεις για τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Εγώ υποστηρίζω την εβδομάδα των 20, την μάλλον περίοδο των 20 εβδομάδων. σχετικά με την άδεια πατρότητας ένας από τους στόχους μας είναι ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι αν πετύχουμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεση αυτή την άποψή μας για την άδεια πατρότητας, αυτό θα είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό για την ισότιμη αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών. Εφόσον πιστεύουμε ότι η άδεια μητρότητας είναι ένα δικαίωμα της γυναίκας και εφόσον θέλουμε να υπάρχουν ισότιμα δικαιώματα ανδρών γυναικών, τότε και η άδεια πατρότητας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη συγκεκριμένη πρόταση οδηγίας, πόσο μάλλον που και το δικαίωμα του παιδιού σε κατάλληλη φροντίδα είναι ένα δικαίωμα το οποίο δεν θα πρέπει να αγνοηθεί εφόσον θέλουμε να ε, δράσουμε πράγματι με αποτελεσματικότητα. Για μια ακόμη φορά λοιπόν υποστηρίζω τις θέσεις της ΕΝΤΙΤ και ελπίζω η έκθεση αυτή να καταλήξει μια προοδευτική έκθεση και το Κοινοβούλιο να ακουστεί. Ένα επιπλέον στοιχείο να σας πληροφορήσω ότι η γνωμοδότηση θα ψηφιστεί από την Επιτροπή Απασχόλησης στις 27 Ιανουαρίου. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πλάμπ. Η κυρία Κώστα έχει το λόγο και μετά η κυρία Τόμσον. θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια διαπίστωση. Το θέμα αυτό δεν αφορά τα έλεγα τη συμφιλίωση των ρόλων ανδρός και γυναικός ή των ρόλων της πατρότητας και της μητρότητας αλλά να το βάλω λίγο πιο φιλοσοφικά ανάμεσα στο υλικό και το πνευματικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το οποίο προστατεύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της μητρότητας και να μην κάνουμε ε, θα έλεγα ένα άλμα προς τα εμπρό σε πολιτισμικό επίπεδο, αλλά σαν νομοθέτες να προχωρήσουμε σχετικά με την κουλτούρα του σεβασμού της ισότητας άνδρα-γυναίκας και στον τομέα της, άδρας, της άδειας μητρότητας και πατρότητας. Νομίζω ότι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε θετική την έκθεση αυτή με ε, συγκεκριμένες προσθήκες γιατί το κείμενο πράγματι μπορεί να θεωρηθεί κάπως περιορισμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι δευτερεύον και μπορεί να εμπλουτιστεί. Αυτά τα οποία εξέθεσε τις βασικές επιλογές της η κυρία Εστρέλα αφορούν τη νομική βάση. Υπάρχει μια σαφής επιλογή σε σχέση με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε, να αναζητήσουμε και εδώ ελπίζω η Ισπανική Προεδρία που επέρχεται να βοηθήσει έτσι ώστε να διευρυνθεί η νομική βάση και το περιεχόμενο κατά συνέπεια της οδηγίας για να μπορέσουμε να διευρύνουμε την άδεια μητρότητας και στην πατρότητα και στη γονεϊκή άδεια. Υπενθυμίζω ότι έχουν υπάρξει δύο σημαντικές οδηγίες πίσω μας οι οποίες έχουν αλλάξει την ομοθεσία. Υπάρχει η οδηγία του 92 και αυτή του 96 το να προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη μας και τις δύο πλευρές που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν και να συνδυάζονται την καινούργια αυτή οδηγία, νομίζω ότι είναι κάτι το αρκετά υπεύθυνο, είναι ταυτόχρονα ένα βήμα πολιτισμού. Θα εμείνω περισσότερο σε δύο θέματα. Πρώτο, το αναγκαστικό ή όχι, ο όρος αναγκαστικό ο υποχρεωτικός αναγκαστικός χαρακτήρας, κάποιος το είπε ότι έχει ιστορικές καταβολές. Νομίζω ότι η πολιτική μας ιστορία σε όλες σχεδόν τις χώρες είναι ένας τρόπος προστασίας ορισμένων θεμελιωδών στοιχείων. Η προστασία της υγείας της μητέρας, σαν παράδειγμα, η οποία λίγο πριν και μετά τον τοκετό είναι σε στάδιο, θα έλεγα, ιδιαίτερη, ε, είναι, είναι ε, γενικά πολύ ευαίσθητη γυναίκα πριν και μετά τον τοκετό, ευάλωτη πράγματι. Επίσης και προστασία των εργασιακών της δικαιωμάτων, να μην απολύεται, να μην γενικά αντιμετωπίζεται με κατώτερο τρόπο Εγώ λοιπόν δεν είμαι κατά τον υπο, του υποχρεωτικού χαρακτήρα που αφορά αποκλειστικά την γυναίκα, γιατί αυτό αφορά δύο ευάλωτα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την γυναίκα πριν και μετά τον τοκετό. Αν και συμφωνώ βέβαια στο ότι θα πρέπει να προβλέψουμε παράλληλα με το δικαίωμα της γυναίκας, το οποίο είναι υποχρεωτικό θα έλεγα σαν φροντίδα γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είναι θέμα επιλογής αλλά είναι ένα θέμα θα έλεγα προστασίας του προσώπου από την κοινωνική και εργασιακή συγκυρία. Θα πρέπει λοιπόν παράλληλα με αυτό το δικαίωμα να υπάρχει επίσης ένα προστατευόμενο δικαίωμα και όχι εδώ κάτι το υποχρεωτικό και αναγκαστικό του πατέρα να μπορεί Κατά τη διάρκεια αυτής της λεγόμενης ε, υποχρεωτικής περίοδου στην Ιταλία είναι δύο μήνες συν τρεις ή τρεις μήνες μάλλον συν δύο να εξελίσσεται παράλληλα και αυτό το δικαίωμα για τον πατέρα να έχει δικαίωμα στην πλήρη πληρωμή να αμείβεται κανονικά εφόσον δεν αμείβεται εν πάση περιπτώσει ειδικά ο πατέρας αυτό θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά για τη μητέρα αν και η μητέρα συνήθως έχει χαμηλότερες αμοιβέ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει το δικαίωμα για την αμοιβή την πλήρη και για τον άνδρα και έχει μεγάλη σημασία να υπογραμμίσουμε επίσης και κάποιες ε, και ε, καινοτομίες, ε, ένα παιδί το οποίο ας πούμε μετά από υιοθεσία μπαίνει σε μια οικογένεια, είναι ουσιαστικά μια νέα γένα για την οικογένεια αυτή. Οπότε θα πρέπει εδώ να ε, υπάρχει η ίδια μορφή κάλυψης και προστασίας των οικογενειακών δικαιωμάτων. Η αρχή της επικουρικότητας, η οποία δεν υπογραμμίζεται πάρα πολύ, λέγεται βέβαια ότι καλούνται τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό, καλούνται τα κράτη-μέλη να κάνουν εκείνο. Πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα μάλλον και το καθήκον των κρατών μελών και να προσαρμοστούν και να προωθήσουν τις θέσεις της οδηγίας και θα πρέπει και η εθνική νομοθεσία να αλλάξει εκεί όπου είναι πιο πίσω από την κοινοτική νομοθεσία ή το αντίθετο και σε σχέση με αυτά τα οποία έλεγε η κυρία Λουλούλινγκ ότι θα πρέπει δηλαδή τα θέματα που ισχύουν για τον άνδρα και τη γυναίκα να εκφραστούν με διαφορετικό τρόπο. Όχι, εδώ θα πρέπει το Κοινοβούλιο να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός. Θα πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν με μια ολοκληρωμένο τρόπο αυτό το οποίο ίσως ε, να μην είναι κοινό σε όλους, ο τρόπος δηλαδή που χορηγείται η άδεια μητρότητας, η άδεια πατρότητας και η γονεϊκή άδεια. Το θέμα εδώ είναι να το δούμε συνολικά, το θέμα είναι να το δούμε σφαιρικά όπως πολλές φορές τίθεται και ε, με φιλοσοφικό τρόπο αν θέλετε και το θέμα της επιμέρους απασχόλησης ε, κατά τη διάρκεια της εργασιακής ζωής. Πρέπει λοιπόν με πολύ συνολικότερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα των τριών τύπων άδειας που παίρνουν οι γονείς. Λοιπόν, όλο το κοινοβούλιο πρέπει να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός. Αυτό θα είναι καλό και για τις γυναίκες και για τους άνδρες. Είναι μια ειδική μέρα σήμερα η 1η Δεκεμβρίου και καλό θα είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα πεδίο συνεννόησης μέσω τροπολόγησης και όχι απόρριψης κάποιων στοιχείων τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θεωρούν αρνητικά και απαράδεκτα οι γυναίκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζοντας όμως ότι οι τελευταίες οδηγίες, η τελευταία είναι εδώ και 13 χρόνια, οπότε προφανώς έχει έρθει η ώρα να κάνουμε ένα προς τα εμπρός βήμα. Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Η ε, κυρία σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ιόβια υπομονή που έδειξε κατά την εκπόνηση της έκθεσης. Είναι πολύ σημαντικό να επιμείνετε στα θέματα αρχής και για την άδεια πατρότητας. Θα πρέπει να δικαιούνται και οι πατέρες να λαμβάνουν άδεια. Χθε ακούσαμε τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μισθολογικό χάσμα και τη διαφορά των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Η πιο σοβαρή διαφορά στις αμοιβέ αρχίζει με την τεκνοπία, γιατί τότε οι άνδρες εργάζονται περισσότερο, οι γυναίκες λιγότερο και οι θέσεις α, τις οποίες διεκδικούν δυστυχώς είναι χειρότερης ποιότητας. Και αυτή η κατάσταση αντανακλάται και στην οικογένεια. Γι' αυτό η πρόταση αυτή είναι το πρώτο βήμα αποκατάστασης μη ισορροπίας. Όταν ε, μιλούν ομοειδεάτες για τα θέματα ισότητας και για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λένε ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε την ισότητα, αλλά δεν πρέπει οι γυναίκες να έχουν το μονοπόλιο στην ανατροφή των παιδιών, θα πρέπει και εμείς οι πατέρες ε, να συμμετέχουμε σε αυτήν και να δικαιούμαστε άδεια πατρότητας. Νομίζω ότι εκεί είναι κοινό ο στόχος και με τους άνδρες. Η οδηγία βέβαια εδράζεται στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή και ήδη πολλές φορές μέλη έχουν ήδη θεσμοθετημένη την ε, άδεια πατρότητας δύο εβδομάδων. Στη Δανία, για παράδειγμα, όταν ε, έκανα το παιδί μου και τις πρώτες δύο εβδομάδες είχα και την αρρωγή του σύζυγου μου, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Όλοι, όλες οι γυναίκες λένε ότι όταν επιστρέφουν από, τη, από το μεευτήριο θέλουν να, έχουν τη συμπαράσταση και την έμπρακτη βοήθεια από τους σύζυγους τους. Γιατί είναι πολύ ευάλωτοι η μητέρα τις πρώτες εβδομάδες αμέσως μετά το κετό και εκείνη που μπορεί να συνδράμει ιδιαίτερα ο πατέρας. Νομίζω όμως ότι η πρότασή μας θα πρέπει να αλλοιώνει τις προτάσεις αυτές και να ισοπεδώνει προς τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Για παράδειγμα, στην Ισπανία η άδεια πατρότητας είναι τέσσερις εβδομάδες. Γιατί να εναρμονιζόμαστε προς τα κάτω. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές νοοτροπίες, αλλά αυτή είναι η προσφορά, είναι δικαίωμα. Δεν θα τιμωρηθεί ο πατέρας που δεν αξιοποιεί αυτό το δικαίωμα των δύο εβδομάδων, αλλά να μπορεί τουλάχιστον να έχει αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστούμε κύριε Τόμσον και κύριο Σιμάνσκι. Κυρία Πρόεδρε, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και την ακούω με κάποια σύγχυση και με μία μικρή θλίψη, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα ήταν πολύ αρνητικό η έκθεσή μας και η θέση μας να περάσει με πλειοψηφία ή να απορριφθεί. Νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό το θέμα που η Επιτροπή μας θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να καταλήξει συνένεση και να μην περάσει με απλή πλειοψηφία να περάσει έκθεση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση ως προς την άδεια πατρότητα, την άδεια μητρότητα, στη γονική άδεια. Η διαφορά είναι ως προς τη μορφή και τον χώρο που θα ε, περιλάβω αυτά τα θέματα. Το θέμα είναι οι προτάσεις θα ενισχύσουν αυτή την κατάσταση ή θα την αποδυναμώσουν. Θα βάλουν κάποια τάξη ή θα δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες διαφορές. Γιατί μερικές φορές ε, έχουμε κάποιες ε, παραδοσιακές ε, συντηρητικές απόψεις ότι αυτές οι άδειες είναι Απόπειρε ανατροπή του παραδοσιακού οικογενειακού μοντέλου. Ενώ αντίθετα η άλλη πλευρά ε, θεωρεί ότι έτσι απαξιώνεται ο πατέρας. Κάποιος όμως πατέρας, ε, εγώ ως πατέρας που έχει πέντε παιδιά, επαναλαμβάνω την εμπειρία μου ότι και ο πατέρας θα πρέπει να βοηθήσει τη μητέρα, θα πρέπει να είναι παρόν στο σπίτι, να, την, να τη συμπαρασταθεί, να συνδράμει. Αλλά δυστυχώς και Εκατό χρόνια να εργαζόμαστε στο σημείο αυτό. Αποκλείεται ο πατέρα να αντικαταστήσει τη μητέρα. Και εγώ έβγαλα όλα τα παιδιά μου, τα έκανα μπάνιο, τα, τα έθρεψα, αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να υποκαταστήσω την γυναίκα μου στο θυλασμό. Και πραγματικά ε, αισθανόμαστε μερικέ φορέ ανήμποροι απέναντι στα παιδιά. Και σίγουρα όταν έπαιρνα το παιδί στα χέρια μου ε, είχε, έδειχνε χαρά, αλλά όταν το έπιανε η μάνα στην αγκαλιά της έδειχνε πραγματική ευτυχία, ευδαιμονία. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ενδώσουμε σε μια συγκινησιακή συζήτηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πρώτα απ' όλα τα συμφέροντα των ανδρών και των γυναικών. Και σίγουρα η Σουηδία έχει πολύ διαφορετική άποψη από τις άλλες χώρες. Αν δεν υπάρχει άδεια μητρότητας, υποχρεωτική για κάποιες εβδομάδες, τότε η κατάσταση που αναφέραμε χθε θα επαναληφθεί. Γιατί ήδη είναι δύσκολη η κατάσταση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και ο εργοδότης ήδη τον προσλαμβάνει μια γυναίκα, τη ρωτάει για την προθέση της, αν θα μείνει έγκυος, αν θα κάνει παιδιά. Αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά δυστυχώς τέτοιες πρακτικές εφαρμόζονται. Αν όμως δεν υπάρχει υποχρεωτική άδεια μητρότητα ή και άδεια πατρότητα, τέτοιου είδους καταστάσεις θα τις εκμεταλλευτούν οι εργοδότες. αρκεί και μία υπόθεση ε, και γυναίκα που δεν έχει χέγγια για την υποχρεωτική μητρότητα σίγουρα δεν θα ασκήσει το δικαίωμά τη αν φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά τη. Νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό το σημείο και αυτό σα το λέει κάποιο από μια χώρα που πρόσφατα προσχώρησε στην Ένωση. Επίση, θα πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα όχι υπό το πρίσμα μόνο του εργοδότη, του εργαζόμενου, τη ε, μητέρα ή του πατέρα, αλλά και από το πρίσμα των παιδιών. Και μάλιστα η έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας λέει ότι η προστασία της μητρότητας ε, εξυπηρετεί κυρίως το συμφέρον των παιδιών. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη και να μην το ξεχνούμε. Επίσης να μην είμαστε αφελείς και να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Ε, πολλές φορές ε, οι επικρίσεις και οι οφείλονται στα οικονομικά ζητήματα. Γιατί το κεφάλαιο και τα συμφέροντα των ε, επιχειρηματιών φυσικά είναι κατά της μητρότητας, γιατί δεν θέλουν να στερούνται την εργαζόμενη για ένα διάστημα. Αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η δική μας Επιτροπή θα, δώσει, θα πρέπει να δώσουμε μάχη υπέρ των γυναικών και υπέρ της μητρότητας και να είμαστε κατηγορηματικοί και επίμονοι. Πολλές φορές το θέμα είναι οικονομικό, αλλά δυστυχώς ακόμη και οι εγγύσεις που δίνουν τα κράτη είναι πολύ διαφορετικέ. Γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια εναρμόνιση. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να σταθούμε ένα λεπτό και να προβληματιστούμε και να δούμε τι διατύπωση θα υιοθετήσουμε, γιατί και ο τίτλος είναι περιοριστικός που μιλά για έγκυες, λεχόνες, γαλουχούσες, αλλά αναφερόμαστε και σε άλλα θέματα. Αυτό όμως δημιουργεί μια σύγχυση, για να μην, έλεγα, για να μην πω χάος, και μια σημαντική διαφοροποίηση. Και ίσως μια τέτοια διάσπαση έχει το αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Θα ήθελα να σε απευθύνω έκκληση. Μήπως θα πρέπει να προβλέψουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε καλύτερα τα πράγματα αυτά. Γιατί και το θέμα της οδηγίας πατρότητας ε, είναι σημαντική και ίσως αν έχει το χαρακτήρα οδηγίας ε, θα εξασφαλίσει κάποιες εγγύσεις. Μήπως δεν θα πρέπει να επιφέρουμε αναγκαστικά μια τέτοια έκθεση, αλλά να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε για περισσότερο χρόνο ποια είναι η κατάλληλη λύση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας θυμίζω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, γιατί η κυρία Εστρέλα πρέπει να φύγει στις 11. Εγώ δεν θα ξαναπάρω το λόγο. Κυρία Ζαμπόρσκα παρακαλώ να είστε σχετικά σύντομοι γιατί θα ήθελα να δώσω το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο τέλος στην εισηγήτρια. Ζαμπόρσκα. E, Κοιτάξτε, ήθελα απλά να πω το εξή για να, ε, να το πω τώρα για να μην υπάρξουν παρεξηγήσει στο μέλλον. Το ΕΛΚ στηρίζει την άδεια πατρότητας. Στηρίζουμε την ε, οικογενειακή άδεια. Επιθυμούμε και οι πατέρες να αναλαμβάνουν την μέρημνα των παιδιών. Και αν δείτε λιγάκι τις ε, εκθέσεις μου, θα διαπιστώσετε ότι σε όλες μου τις εκθέσεις ε, ομιλώ για την μέρημνα του πατέρα για τα παιδιά. Όμως ένα πράγμα δεν επιθυμούμε. Σε αυτή την οδηγία όπου γίνεται λόγος για την υγεία της ε, μητέρας δεν θέλω να υπάρξει εξίσωση και των τριών δυνατοτήτων άδεια. Δηλαδή υπάρχουν οι εξή λύσει. Είτε θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, όμω θα παραμείνουμε αυστηρά προσκολλημένοι στου όρου οδηγίε. Αυτή είναι μία δυνατότητα. Η άλλη δυνατότητα που υπάρχει είναι να μα δοθούν και τα τρία κείμενα της Επιτροπής και μετά να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Υπάρχει μια τρίτη δυνατότητα, αν όλοι συμφωνούμε, να υποβάλουμε μια συγκεκριμένη ερώτηση προς την Κομισιόν, έτσι ώστε η Κομισιόν να προετοιμάσει και αυτή συγκεκριμένο έγγραφο, όπου θα αναφέρονται σε ένα και μόνο έγγραφο και τα τρία είδη της ε, άδεια. Ευχαριστούμε κυρία Ζεμπόφσκα. Η Κομισιόν λοιπόν τώρα θα λάβει το λόγο. Νομίζω ο κύριος Ούλσον είναι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι, σύντομος. Και να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Εστρέλα και όλους τους άλλους που συνέβαλαν ε, σε, αυτό το, σε αυτή τη συζήτηση. Βρήκα τη συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα καθότι αντικατοπτρίζει και την περίπλοκη μορφή αλλά και τη σημασία της ε, συνδιαλλαγής η οποία οποία ε, χαρακτηρίστηκε από όλε αυτές ε, τις ε, μορφές αδειών που υπάρχουν και τα δημογραφικά θέματα που βεβαίω όλα πρέπει να εξεταστούν συνδυασμένα. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που σας παρουσιάστηκαν εχθές για τα θέματα που συζητάμε. η συνάδελφός μου και εγώ ήρθαμε απλά σήμερα εδώ για να διευκνήσουμε τεχνικής φύσεως θέματα. Ε, γνωρίζετε ότι η Κομισιόν ε, αυτή τη στιγμή ε, είναι μεταβατική αν θέλετε με αυτή την έννοια. Σύντομα θα αναλάβει νέος επίτροπος για τις δικές μας αρμοδιότητες και τότε θα διαμορφωθεί και η τελική θέση για την έκθεση. Βεβαίως ο Επίτροπος κύριος ε, Σπίντλα και το Σώμα των Επιτρόπων έχουν ήδη τοποθετηθεί σε πάρα πολλά θέματα. Εγώ δεν θέλω να τα επαναλάβω αυτά. Υπάρχουν ε, στη διάθεσή σας, δεν θέλω να χρονοτριβήσω από αυτόν. Τώρα, κάποιες διευκρινήσεις. Ε, το Συμβούλιο κοινωνικών υποθέσεων και ίσων ευκαιριών ε, συνήλθε εχθές ε, και συμφώνησε για την οδηγία περί γονεϊκής άδειας. Άρα δηλαδή έχουμε την πολιτική συμφωνία για αυτή τη μορφή άδεια, τη γονεϊκή άδεια, η οποία χορηγεί το δικαίωμα σε κάθε ένα από τους δύο γονείς ε, τεσσάρων μηνών άδειας. Και υπάρχει και μια άλλη καινοτομία, ένας μήνας που δεν μεταφέρεται Δηλαδή τι σημαίνει αυτό κύριε Πρόεδρε. Σημαίνει de facto ότι αν ο πατέρας δεν ε, κάνει χρήση αυτού δικαιώματος ε, του ενός μήνος άδεια, το δικαίωμα αυτό χάνεται. Δεν μπορεί να μεταφερθεί. Δεύτερον, εχθές το Συμβούλιο κατέληξε και σε άλλη πολιτική συμφωνία σχετικά με τους αυτοπασχολούμενους ε, και την ε, σχετική οδηγία που αφορά την αρρωγή στις ε, συζύγους τους. Υπάρχει πολιτική απόφαση ότι το θέμα αυτό θα συνεχιστεί υπό την Ισπανική Προεδρία για τη δεύτερη ανάγνωση. Τρίτον, όσον αφορά την άδεια πατρότητα, α είμαστε σαφεί. Αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσει επί του θέματο. Η Επιτροπή ανακοίνωσε με απόλυτη σαφήνεια ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο και ξεκινάμε βασιζόμενοι στη χθεσινή συμφωνία, στη χθεσινή οδηγία για την ε, άδεια πατρότητας και ξεκινάμε και θα προβούμε σε ενδελεχή οικονομική ανάλυση της κατάστασης. Θα προετοιμάσουμε μελέτη αντικτύπου για το θέμα αυτό και τέλος η, απόφαση, ε, η πολιτική απόφαση θα ληφθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση επί του θέματος και ούτε πρόκειται να ληφθεί απόφαση αμέσως επόμενους μήνες. Όπως σας είπα για την ε, άδεια πατρότητα. Ε, η Επιτροπή τοποθετήθηκε από αυτού το Μάιο, αλλά θα ήθελα να αναφέρω κάποια θέματα που τα κρίνω σημαντικά. Η έκθεση αυτή ενισχύει την ευελιξία με την έννοια ότι προβλέπει το δικαίωμα για τη μητέρα να κάνει χρήση της γονεϊκής άδεια. Άρα δηλαδή κράτη-μέλη που έχουν πολύ γενναιόδορες ρυθμίσεις για τη γονεϊκή άδεια, αυτά τα κράτη μπορούν να συνυπολογίσουν αυτή τη γονική άδεια μέσα στην άδεια μητρότητας που θα αποφασιστεί από το Σώμα των Επιτρόπων. Και αυτή είναι μια σημαντική προσθήκη με την έννοια ότι το θέμα αυτό είχε προκαλέσει κάποιες επιφυλάξεις στο Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν τελικά πρόκειται για ένα θέμα ε, επί του οποίου θα μπορούσε στο μέλλον να υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο. Άρα δηλαδή αν θέλετε αυτή είναι μια θετική προσθήκη ή διευκρίνηση στην έκθεση. Και άλλο ένα θέμα τεχνικής φύσεως, ότι πρόκειται μια οδηγία που εμπίπτει στην οδηγία πλαίσιο περί υγείας και ασφάλειας, η οποία προβλέπει και αλλο ενα θεμα τεχνικη φύσεω, οτι προκειται μια οδηγια που εμπιπτει στην οδηγια πλαισιο περι υγειας και ασφαλεια η οποια προβλεπει και τεχνικου ε, περιορισμου ε, για το πεδίο εφαρμογή και άλλα παρεμφερή θέματα. Υπάρχει μια προσθήκη για οικιακού ε, ή οικιακέ βοηθούς. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ρυθμιστεί στην οδηγία πλαίσιο και όχι στην ειδική οδηγία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτέ είναι οδηγίε που μπορώ να σας τι ε, ε, διευκρινήσει μπορώ να σας απαντήσω, να σας δώσω και κατηδίαν και να μην σπαταλάμε το χρόνο των υπολείπων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ε, κυρία Στρέλλα, η συγκεκριά μας, έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για αυτή την πολύ γόνιμη και ζωντανή συζήτηση. Πολύ ζωηρή αυτή η συζήτηση στην οποία συμμετείχε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που μας έδωσε πολύ χρήσιμες πληροφορίες στο τέλος. Θα είμαι επιγραμματική γιατί όπως σας είπα και στην αρχή θα φύγω για την Λισαβόνα και σίγουρα <laughs> δεν θα με περιμένει το αεροπλάνο να καθυστερήσω. Σε γενικές γραμμές λοιπόν και κρίμα που έφυγε η κυρία Λούλη δεν πρόκειται να της απαντήσω εκτενώς. Θα ήθελα πάντως να τη διαβεβαιώσω ότι παίρνω πολύ στα σοβαρά το έργο μου και όχι μόνο το δικό μου αλλά και της Επιτροπής μας. Και αν υπάρχουν κάποιοι που δεν παίρνουν στα σοβαρά είτε τον εαυτό τους είτε το έργο των άλλων είναι δικό τους πρόβλημα. Άλλωστε υπήρξαν εξελίξεις, παρακολουθούμε τις εξελίξεις των καιρών. Δεν μείναμε ε, ακινητοποιημένοι στο χρόνο, δεν ε, έχουμε παραλύσει στην έκθεση και την κατάσταση του 1966. Υπήρξαν κάποιε παρεξηγήσεις Εγώ δεν μιλώ για τη γονική άδεια. Μιλώ μόνο για την άδεια μητρότητας και την άδεια πατρότητας Και γνωρίζω ότι σε μερικές γλώσσες η μετάφραση μπορεί να δημιουργήσει παρανοήσει. Θα ήθελα όμως να διευκρινίσω ότι έχουμε μια οδηγία που αναφέρεται στη γονική άδεια και που τη διαπραγματευτήκαμε με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά δεν θα περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η οδηγία για τη γονική άδεια δεν θα περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έχουμε άλλη οδηγία για την άδεια μητρότητας, που είναι αυτή που αναθεωρούμε τώρα. Και κατά τη γνώμη μου, αλλά και κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων, με εξαίρεση ίσως το ΕΛΚ και του κ. Σιμάσκη, συμπεριέλαβα και την άδεια πατρότητα στην έκθεσή μου, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα δικαιώματα είναι θεμελιώδη και συμπληρωματικά. Και φυσικά η αντιπατρότητα δεν αναφέρεται σε μια περίοδο που η μητέρα είναι αναντικατάσταση, αναντικατάστατη. Αλλά σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, στους πρώτους έξι μήνες η γυναίκα ανακάμπτει. Αλλά μέσα αυτό το διάστημα μπορεί να γίνει ένας επιμερισμό των οικογενειακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αλλά και για το παιδί το παιδί έχει δικαίωμα να έχει στο σπίτι και, το, και τη μητέρα του και τον πατέρα του και χρειάζεται την βοήθεια και τη στήριξη και των δύο. Και η οικογένεια έχει δικαίωμα σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή να είναι ενωμένη, να μοιράζονται οι δύο σύντροφοι τις ευθύνες, να μοιράζονται την μοναδική αυτή χαρά και αυτή τη μοναδική στιγμή στον οικογενειακό τους βίο. Μάλιστα 17 χώρες μέλη ήδη έχουν κατοχυρώσει την άδεια πατρότητας. 17 κράτη-μέλη επαναλαμβάνω. Εγώ αυτό που προσπάθησα είναι να προσαρμόσω την κατάσταση που ήδη ισχύει σε πολλά κράτη-μέλη και να ενθαρρύνω και τις υπόλοιπες χώρες να μιμηθούν το παράδειγμα των πιο προοδευτικών νομοθεσιών και να κατοχυρώσουν και αυτές την άδεια πατρότητας. Και σας είπα ότι είμαι απόλυτα ε, ανοιχτή και διαλλακτική για να βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Θα εργαστούμε με σοβαρότητα και χωρίς προκαταλήψεις. Σίγουρα καμία λέξη δεν είναι ουδέτερη ή ανώδυνη όλες οι λέξεις έχουν το νόημά τους και ίσως διαφορετικό βάρος σε κάθε χώρα. Γι' αυτό και απέσυρα το χαρακτηρισμό υποχρεωτική από την άδεια πατρότητας, ύστερα από αίτημα των φιλελευθέρων. Γιατί κατά τη γνώμη των φιλελευθέρων, ο όρος υποχρεωτικός ε, έχει ιδιαίτερο βάρος και γι' αυτό απέσυρα το υποχρεωτικό από την άδεια πατρότητας. Για να σας δείξω πόσο διαλεκτική μου και πόσες ε, προτάσεις ενσωμάτωσα. Και λυπούμε που το ΕΛΚ δεν έστειλε τις αντιρρήσεις ή τις παρατηρήσεις ή τις επικρίσεις και τις τροπολογίες του για να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Γιατί τι νόημα έχει στη διάρκεια της συζήτησης να μας εκθέτει το ΕΛΚ τις απόψεις του και τις αντιρρήσεις του. Έπρεπε να είχαν υποβάλει τα σημεία με τα οποία συμφωνούσαν, αυτά με τα οποία διαφωνούσαν και τις προτάσεις για να συνεργαστούμε. Εγώ θέλω να συνεργαστώ και με το ΕΛΚ. Γιατί το ΕΛΚ είναι μια πολύ σημαντική πολιτική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να μου πει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πού έγινε οι βασικές αντιρρήσεις του. Τι αισθάσεις έχει το ΕΛΚ με την έκθεση. Θα έχουμε και νέο επίτροπο αρμόδιο για θέματα ισότητας. Θα έχουμε και νέα προεδρία σε λίγο. Θα συνεργαστούμε λοιπόν και με την επόμενη προεδρία για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Θα ήθελα εν τέλει να ευχαριστήσω θερμά την ε, κυρία Ροβάνα Πλάμ, που είναι η συγγήτρια της γνωμοδότησης από την Επιτροπή Απασχόλησης. Είχαμε πολύ στενή και αγαστή συνεργασία και προσπαθήσαμε να συμβάσουμε τις απόψεις μας. Σας ευχαριστώ και λυπούμε που θα φύγω κάπως εσπευσμένα, αλλά είναι για καλό σκοπό γιατί θέλω να είμαι στη Λισαβόνα κατά την πανηγυρική στιγμή έναρξης της εφαρμογής της συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στρέλα. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ όλους ε, τους ε, συναδέλφους, ε, γιατί η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Άλλοι τέσσερις ε, ε, είχαν ζητήσει το λόγο για να κάνουν τις ε, παρεμβάσεις τους. Κυρία Στρέλα πρέπει να φύγει. Αν θέλουν όμως οι τέσσερις αυτοί μπορούν να μιλήσουν τώρα. Παραδείγματο χάρη ο κύριος Ρουμέβα είχε ζητήσει το λόγο, η κυρία Μπάουα και αν θέλετε να κάνετε κάποιες σύντομες παρατηρήσεις θα σας δοθεί η δυνατότητα. Πάντως η κυρία Στρέλα πραγματικά πρέπει να φύγει τώρα. Πριν λοιπόν φύγει η κυρία Στρέλα, θα ήθελα να πω ότι ε, στις 15 Δεκεμβρίου εκπνέει στις 12 το μεσημέρι η τελική προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Και ε, θα συμφωνήσουμε, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 23 Φεβρουαρίου και όλο το θέμα θα παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του ε, Μαρτίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Στρέλα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Ρωμέβα θέλει τώρα να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Θα ήθελα να υποστηρίξω την γραμμή της εισηγήτριας. Λυπούμε που έφτασα καθυστερημένα, αλλά εστερνίζομαι αυτά που μας είπε η εισηγήτρια κυρία Στρελακή για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της άδειας πατρότης, που είναι κάτι που θα επαναλάβουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ και θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Η κυρία Μπάουερ είχε ένα νέο σχόλιο. Κοιτάξτε, λυπάμαι πάρα πολύ για το ότι ε, έπρεπε να φύγει η κυρία Στρέλα. Εγώ ε, ήθελα να της πω το εξής ε, προσπάθησε να βγάλει αυτή την υποχρεωτική ε, διατύπωση αλλά στο 16 εξακολουθεί να αναφέρεται και το άρθρο αυτό ε, καθιστά σαφές ότι όσα κρατημέλη δεν έχουν ήδη εισάγει αυτή την διατύπωση υποχρεούνται να το πράξουν σχετικά με την άδεια πατρότητα. Δεν ξέρω πώς δεν το πρόσεξε αυτό η κυρία Εστρέλα. Θέλω όμως να πω το εξή ε, και λυπάμαι πάρα πολύ που έπρεπε να φύγει η κυρία Εστρέλα. Το θέμα δεν είναι ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι κατά ε, της ε, άδειας πατρότητας ή της ε, οικογενειακής άδειας. Δεν θέλουμε εμείς να καθορίσουμε το τι θα περιλαμβάνει η οδηγία. Θέλουμε μόνο να καταθέσουμε μια πρόταση να υπάρχει μια σύγχρονη πρόταση και γι' αυτό λοιπόν επιθυμούμε να επιμείνουμε στο ότι η οδηγία αυτή πρέπει να παραμείνει ως οδηγία ασφάλειας και υγείας. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που παραπέμπουν ε, στο ότι χρειαζόμαστε ε, πιο ευέλικτες ε, μορφές άδειας πατρότητας ή οικογενειακής άδειας δεν πρόκειται όμως μόνο για μία μορφή άδεια. Και σε τελική ανάλυση δεν έχει κανένα νόημα να προσθέσουμε άλλη μία διατύπωση σε αυτές που ήδη υπάρχουν και είναι πολύ καλές. Οι υπερβολικές προτάσεις είναι λάθος. Παραδείγματο χάνει το θέμα της διάστασης του φύλου, το mainstreaming. Άτοπο, δεν έχει καμία σχέση και στην ε, άδεια πατρότητας. Εκεί η άδεια πατρότητα δεν έχει καμία σχέση με το mainstreaming. Βέβαια αυτή ίσως να είναι και η μόνη εξαίρεση. Οι μητέρες πρέπει να προστατευθούν όταν επανέρχονται στην αγορά εργασίας. Το έγγραφο λοιπόν περιλαμβάνει πολυάριθμες, ε, πολύ καλές ε, προτάσεις, όμως ε, το έγγραφο αυτό βρήθη προτάσεων οι οποίες έχουν κατατεθεί καλή την πίστη. Βεβαίως οι προτάσεις αυτές έχουν κατακλείσει το έγγραφο, είναι υπερβολικά πολλές και εμείς δεν είχαμε κατά νου να επικρίνουμε την πρόταση των κοινωνικών εταίρων για την άδεια πατρότητας. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Υπάρχουν στο έγγραφο και άτοπες παρατηρήσεις, προτάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το έγγραφο και αλλοιώνουν το νόημα και την ουσία. Εξ όσων λοιπόν γνωρίζω και η ε, Επιτροπή σκέπτεται ότι αν τελικά το έγγραφο αυτό εγκριθεί θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν οι διατάξεις του. Οι μητέρες ε, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση έτσι κι αλλιώς και δεν χρειάζονται προστασία που είναι ανεφάρμοστη. Αυτή είναι η μόνη διαφορά που υπάρχει ανάμεσά μας. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μέχρι οι κοινωνικοί εταίροι να συμφωνήσουν για την άδεια πατρότητας. Στο πρόγραμμα εργασίας υπήρχε αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Στρέλα λοιπόν συμπεριέλαβε ε, το θέμα της άδεια απατρότητας σε αυτή την πρόταση οδηγίας και με τον τρόπο αυτό ε, μόνοι μας ε, κάνουμε δύσκολη τη ζωή μας. Δεν θέλουμε να πειράσουμε τη συμφωνία ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν πρέπει να προτρέξουμε. Πρόκειται για μέθοδο και για το ερώτημα τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η οδηγία και τι ενδεχομένως κάποια άλλη. Αλλά για να καταλήξουμε στην άλλη χρειαζόμαστε χρόνο. Και δεν πρέπει βεβαιασμένα να τα ε, συμπιέσουμε όλα σε μία και μόνο οδηγία ή σε μία και μόνο πρόταση. Γιατί με τον τρόπο αυτό η κατανόηση ε, αλλά και η εφαρμογή καθίστανται πάρα πολύ δύσκολες. Ελπίζω λοιπόν ότι η κυρία Εστρέλα η... να άφησε εδώ τουλάχιστον τη βοηθό της και θα ήθελα η βοηθός της κυρίας Εστρέλα να κατανοήσει ότι εμείς δεν είναι ότι ε, διαφωνούμε με όλες τις προτάσεις, απλά θέλουμε να επισημάνουμε ότι δεν επιτρέπεται να πλατιάσει το περιεχόμενο. Και πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τις προτάσεις της ε, Κομισιόν ή αν θέλετε την άποψη των κοινωνικών εταίρων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπάουερ. Ναι, πραγματικά είναι κρίμα που δεν μπόρεσε να παραμείνει μέχρι το τέλος της συζήτησης η κυρία Στρέλλα, Γιατί είχα και εγώ κάποια σχόλια που ήθελα να υποβάλω. Αλλά δυστυχώς έφυγε η συγκεκριτή. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να ολοκληρώσουμε εδώ τη συζήτηση και έχετε λάβει τις ε, πληροφορίες ε, για τις τροπολογίες. Θα ήθελα πάντως να σας απευθύνω έκκληση ε, για να είμαστε διαλλακτικοί, ανοιχτόμυαλοι και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τις μητέρες, τους πατέρες αλλά και τα παιδιά στο μέλλον. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο και να περάσουμε στο επόμενο που προβλέπει ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών από την αντιπροσωπεία της Επιτροπής ε, στη Μαδρίτη. Δεκαμελής ήταν η αντιπροσωπεία αυτή που μετέβη στη Μαδρίτη και εκτός ποσοστώσεως και συμμετείχαν εκεί μέλη της γραμματείας, των πολιτικών ομάδων. βασικός στόχος του ταξιδιού αυτού ήταν να προετοιμάσουμε την επερχόμενη Ισπανική Προεδρία και να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις για το πώς αντιμετωπίζει η Ισπανία τα θέματα ισότητας των δύο φύλων. Και ήδη θελήσαμε να εγκαινιάσουμε τις επαφές μας με την Ισπανική Προεδρία ώστε να έχουμε αγαστή συνεργασία και στη διάρκεια της Ισπανικής αυτής Προεδρίας. Συναντηθήκαμε ε, με την Υπουργό Ισότητας. Παρακαλώ λίγο ησυχία γιατί γίνεται μεγάλη φασαρία στην αίθουσα. Συναντηθήκαμε λοιπόν με την κυρία Πιμπιάνα Άιντο που είναι η αρμόδια υπουργό για θέματα ισότητας και ενημερωθήκαμε για τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας στα θέματα ισότητας. Η υπουργό αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και δήλωσε ότι η Ισπανική Προεδρία θα προτείνει ένα ευρωπαϊκό μορατόριο για τη βία κατά των γυναικών. Μία άλλη προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας σε θέματα ισότητας είναι το θέμα των συνεπειών της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και της αναθεώρησης της στρατηγικής της Λισαβόνας. και στα θέματα αυτά θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των δύο φύλων. Ένα άλλο θέμα είναι η βία κατά των γυναικών και η ισχύουσα ισπανική νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Συζητήσαμε και το θέμα της εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας στην Ισπανία. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, Μιλήσαμε για την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας, την κατάρτιση, την επιμόρφωση, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, το συνδυασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, συναντηθήκαμε και με τον Υφυπουργό για τα θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Διέγκο Λόπες Γκαρίντο, στη διάρκεια γεύματος εργασίας. Ο κύριος Γκαρίντο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και είπε ότι το θέμα αυτό μαζί με την ενέργεια και την προσπάθεια καταπολέμησης της βίας κατά το γυναικό θα είναι οι ύψιες προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας. Συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους ε, της Βουλής και της Γερουσίας Εκεί συνεχίσαμε τις συζητήσεις για τη βία κατά των γυναικών και για την ισότητα, ιδιαίτερα από οικονομική άποψη και άποψη απασχόλησης. Στη συνέχεια συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο της Μαδρίτης, και τον πρόεδρο και τον νομάρχη και μάλιστα διοργανώθηκε και μια στρογγυλή τράπεζα με συμμετοχή εκπροσώπων ε, της κοινωνίας των πολιτών στην Ισπανία. Εκεί έδωσαν το παρόν πολλές οργανώσεις σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα και κάναμε σημαντικό προπαρασκευαστικό έργο θέτοντας ε, δύο σημαντικά ερωτήματα που θελήσαμε να τα εξετάσουμε με την κοινωνία των πολιτών στην Ισπανία. Για παράδειγμα, ποιε είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε σε θέματα ισότητε και ποιε είναι οι προσδοκίε και οι βασικέ προτεραιότητε τη Ισπανική Προεδρία. Αυτά ήταν τα δύο κεντρικά θέματα ε, τη Τρογγυλή Τράπεζα. Αυτά ήταν εν ολίγης τα στη Μαδρίτη. Ευχαριστώ θερμά τα μέλη που συμμετείχαν στην αποστολή αυτή. Ήταν πολύ χρήσιμη, διαφωτιστική και έγινε μια πολύ γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με την Ισπανική Προεδρία. Κάτι που θα μας βοηθήσει και στη διάρκεια του Ισπανικού εξαμήνου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τη γραμματεία μας που προετοίμασε θαυμάσια αυτό το ταξίδι γιατί έτσι με το διήμερο αυτό εμπλουτίσαμε τις επαφές και τις γνώσεις μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Χιμένες για να την ακούσουμε για την αποστολή αυτή στην Ισπανία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εν συντομία τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας ε, όπως μας εξέθεσε η Υπουργός Μπιμπιάννα Αλμάγρο. Ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της καταπολέμησης ε, της ε, βίας κατά το γενικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το θέμα της απομάκρυνσης των αυτούργων αυτής της βίας, γιατί τέτοια προστασία υπάρχει σε ορισμένες χώρες, αλλά για παράδειγμα, το θύμα μια τέτοια βία μπορεί να προστατεύεται στην Ισπανία, αλλά αν μεταναστεύσει σε άλλη χώρα, μένει ανυπεράσπιστο. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα απομάκρυσης του αυτοργού από το θύμα και να ισχύσει σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Αυτό μας το επισήμανε η Υπουργό και θα είναι ένα θέμα ιδιαίτερα προσφυλέ που θα προσπαθήσει να προωθήσει η Ισπανική Προεδρία το θέμα του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Απομάκρυνση ε, Αυτούργων Βία κατά των γυναικών. Καλώ, σα ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό θέμα με το οποίο ανάμεσα σ' άλλα θα ασχοληθεί η μελλοντική Προεδρία. Πέραν αυτού του παρατηρητηρίου θα πρέπει να υπάρξει ένας πράσινος αριθμός όπως λέμε που να λειτουργεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς Νομίζω ότι μπορέσαμε να εξαντλήσουμε την ημερήσια διάταξη. Είχαμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Νομίζω ότι καταφέραμε να πετύχουμε κάτι σημαντικό. Να ενημερώσουμε ένα τον άλλον ή μία την άλλη για τις θέσεις μας, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πολιτικής μας καταβολής δείχνουμε ότι σε ορισμένα θέματα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους.